Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gestern Abend eine Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. χθε είχαμε μια πολύ καλή συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν αντιμετωπίσαμε και καμία σημαντική δυσκολία μεταξύ των ομάδων. Επομένω, για του χρόνου έχουμε προβλέψει επισκέψει σε ορισμένες πόλεις επί τη ευκαιρία της Πολωνικής Προεδρίας θα πάμε στο Βρότσλαβ. Θα πάμε και στις δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες ε, που δεν έχουν πολύ μία από την άλλη. Δηλαδή στο Τούρκου και το Ταλίν, αλλά αποφασίσαμε να μην πάμε στη Ρώμη, αλλά στο Παλέρμο. Στη Ρώμη είναι εύκολο να πάει κανείς. Το Παλέρμο δεν προσελκύει τόσο πολύ κόσμο. Καλύτερα λοιπόν να πάμε στο Παλέρμο. Νομίζω ότι είναι ένα κενό που πρέπει να το πληρώσουμε. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο Παλέρμο, στη Λισαβόνα και στην Βόρα. Και Υπήρξε πρόταση να παραστούμε στο χειμερινό φεστιβάλ ε, του Σαράκεβο. Η Βοσνία βέβαια δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να μεταβούμε εκεί, θα πρέπει να γίνει αυτό πολύ νωρίς ε, του χρόνου για το χειμερινό φεστιβάλ, όπως είπα. Αλλιώς θα πάμε στην πόλη Εύωρας, που δεν είναι και τόσο γνωστή και είναι πολύ ωραία, αξίζει να πάει κανείς. Για τις τρεις πρώτες λοιπόν μετακινήσεις μας οι αποφάσεις είναι ηλιμένες και μετά θα δούμε αν είναι δυνατό να πάμε στην ε, Βοσνία, αλλιώς θα πάμε στην Εύωρα. Τώρα για την ε, σε αποφάσει των συντονιστών έχουν δημοσιευθεί, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από χθε το βράδυ, αλλά ήθελα να σας τα πω και διαζώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βραβείο Λούξ, έχουμε τις τρει ταινίε ε, για το βραβείο Λούξ που παρουσιάστηκαν ε, στη Βενετία και έχουμε προσκαλέσει τους τρεις ε, σκηνοθέτες Ήταν και οι συνάδελφοι Κώστα Σκούρια, εκτός από εμένα, που στήριξαν και αυτοί αυτή την προσπάθεια. Έχουμε την ταινία η ξένη που ε, είναι γερμανική ταινία και αφορά εγκλήματα τιμής. Έχουμε ένα άλλο φιλμ, ε, Illegal λέγεται, είναι βελγο-λουξεμβούργιο-γαλλική παραγωγή και μια ελληνογερμανική παραγωγή, η Ακαδημία Πλάτωνος, είναι η τρίτη ταινία. Τώρα για το θέμα, πώς να το περιγράψω ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση του να είναι κάποιος ανώτερος από κάποιον άλλο και συγκεκριμένα οι σχέσεις και οι απόψεις των Ελλήνων για τους Αλβανούς που αποκαλύπτεται κάτι μετά, δεν μπορώ να σας το πω όμως τώρα όλο το... Λοιπόν, θα δείξουμε αυτές τις τρεις ταινίε και θα έχουμε την ευκαιρία να τις δούμε τον ε, Οκτώβρη και είναι απαραίτητο να τις δούμε, οπότε σας παρακαλώ ο καθένας τουλάχιστον να φέρει άλλους 10 συναδέλφους να ψηφίσουν γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κοινό του κινηματογράφου και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε την οικονομική του σημασία και μιλάμε για ανθρώπους μεγάλο όνομα στον ε, τομέα αυτών. Λοιπόν, οι ταινίε αυτές, όπως σας είπα, Θεού θέλοντος ε, του χρόνου, εάν το επιτρέψει ο Πρόεδρος, θα τις δείξουμε όχι μόνο εδώ, αλλά και στις πόλεις, στις πρωτεύουσες, στις πρεσβείες σε αντιπροσωπείες σε πάση περιπτώσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί εκεί πέρα να ψηφίσει ο κόσμος. Είναι κάτι το θαυμάσιο αυτό. Έτσι ώστε το Κοινοβούλιο με την πραγματική αυτή επικοινωνία που διηγείται την ευρωπαϊκή ιστορία να μπορέσουμε έτσι να διαφημιστούμε. Αλλά όπως σας είπα, αυτό είναι για του χρόνου. Ήδη φέτος σε πάρα πολλές αντιπροσωπείες, π.χ. στη Γερμανία, στο Βερολίνο και στο Μόναχο, δείχνουν ήδη αυτές τις ταινίε για να υπάρξει έτσι μια προπαρουσίαση. Σκεφτείτε το λοιπόν. Είναι σοβαρή ιστορία, σημαντική υπόθεση και σας παρακαλώ στις ακροάσεις που έχουμε στις 28 Οκτωβρίου θα έρθουν δημιουργοί, θα έρθει ο Wim Wenders που αφιέρωσε το χρόνο του. Α, δεν αν δεν ξέρετε να σας εξηγήσω ποιος είναι. Είναι... Σημαίνει για εμάς πως θα έχουμε μεγάλο αριθμό ακροατών από έξω από το Κοινοβούλιο και θα μιλήσει για τα σημαντικά ζητήματα της διακίνησης των ταινιών. Οπότε νομίζω πως θα έχουμε μια αρκετά καλή ακρόαση η οποία θα βοηθήσει αρκετά αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Είμαστε σε καλό δρόμο. Στο Προεδρείο υπάρχει μια κυρία η οποία εντάξει δεν είναι τόσο φιλική, αλλά νομίζω μπορούμε να την πείσουμε πως δεν είναι πεταμένα λεφτά όπως μας είπε, αλλά είναι ε, κάτι το οποίο μας πάει σε ένα διαφορετικό δρόμο από τα χαρτιά και τα φέγγι βολάν και μας πηγαίνει πιο κοντά στις χαρτιές των ανθρώπων είδαμε όταν πήγαμε και στη Βενετία και συζητήσαμε με τους ε, σκηνοθέτες και είχαμε και την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τα ΜΜΕ, ανακαλύψαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα. Και τέλος, κάτι το οποίο ξέχασα να σας πω, όταν ήμουν στις Κάνες, συναντήθηκα με τους διοργανωτές του Cinema Europa και ε, των ημερών της Βενετίας, ένα κομμάτι του φεστιβάλ της ε, Βενετίας όπου ο προ-προηγούμενος πρόεδρος ο Μπαρσάντη είναι εκεί πέρα πρόεδρος και συμφωνήσαμε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του βραβείου Λούξ να προσκαλέσουμε 27 συνεφίλ από τις 27 χώρες που ήρθαν στη Βενετία, είδανε τις ταινίε, συζήτησαν ο ένας με τον άλλον, δημιουργήθηκε ένα πραγματικό δίκτυο συνεφίλ και θα ήθελα να πω πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο γιατί με τον τρόπο αυτόν ήρθαν νέοι άνθρωποι που δεν θα έρχονταν αλλιώς. Οπότε για πρώτη φορά ακούστηκε νομίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται μόνο ξέρω εγώ, με το ψωμί, το περιβάλλον ή την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και για τον πολιτισμό και ε, με αυτά τα οποία απασχολούν τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, αρκετά με αυτά περνάμε στις υποφορίες. Δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στην ψηφιακή εποχή, το μέλλον του διτού συστήματο του κυρίου Μπέλετ ήταν δύσκολη υπόθεση, αλλά νομίζω πως ο κύριος Μπέλετ τα έκανε όλα και χρειάζεται μόνο να ψηφίσουμε, έτσι. Εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Uh, nur eine Minute. Ένα λεπτάκι μόνο, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αυτό το σχέδιο ψηφίσματος αποτελεί το αντικείμενο ε, πολύ στενών επαφών αν θέλετε με όλους τους ε, εμπλεκομένους, ε, με τους διατηλεπτικούς σταθμούς, με, τα, με τους προσώπους του γραπτού τύπου. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο σε αυτή τη ψηφιακή εποχή, όμως για να παρουσιάσουμε τα πράγματα όσα έχουν θα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα και νομίζω ότι εμείς σαν Ευρωπαίοι πολιτικοί, αν θέλετε, θα πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα, αν θέλετε, για να διατηρήσουμε μια σωστή ισορροπία η οποία είναι κρίσιμη για την δημοκρατία. Γι' αυτό θα ήθελα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους ε, τους κοιόδης ηγητές ε, για την ε, συνεργασία. Σε περισσότερα σημεία του κειμένου καταλήξαμε σε συμφωνία, σε, όχι σε όλα, αλλά τέλος πάντων. Και θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, κυρία Πρόεδρε, γιατί ε, υποστηρίξατε την πρόταση για την έκθεση. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή 88 υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 393 υπέρ κατά αποχές δεκτή 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή 119 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 133 υπέρ κατά ξανά 133 υπέρ να μετρήσουμε κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ αποχές δεκτή 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή 139 υπέρ κατά αποχές δεκτή 141 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3. von Schacke. 3 σχάκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εννέα συμβιβαστική υπέρ. Τι θέλατε. Να ελέγξουμε. Εάν δεν έχετε την κάρτα σας να μετρήσουμε. No? Okay, then we, then we check it like this. Okay, we, we check it and then we count the others. Okay. Θα επαληθεύσουμε και μετά θα μετρήσουμε τους υπόλοιπους. Ποιος είναι υπέρ της... Άρχεται η ψηφοφορία μάλλον, συγγνώμη. Η Πέρας. 14 κατά, 9 υπέρ. Μαρία, τι, Μαρία, τι ψηφίζεις. Υπέρ ή κατά. Α, έχεις ψήφισες με την κάρτα. Α, εντάξει, εντάξει, όλα ωραία. Και εσείς είστε υπέρ, κατά. Κατά. Και εσείς κατά. 17 κατά, 9 υπέρ. Μάλιστα, απορρίπτεται, ευχαριστώ. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά εποχές δεκτή 18 καταπίπτει 20 υπέρ κατά εποχές δεκτή συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά να πρέπει να επαληθεύσουμε 43 του εισηγητή υπέρ παρακαλώ ψηλά τα χέρια κατά μάλιστα δεκτή συμβαστική 15 υπέρ δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ 40 κατά με συγχωρείτε αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 απορρίπτεται συγγνώμη σαν τον κύριο Πιτέλα την έχω πάθει. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 όχι 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην τελική ψηφοφορία να γίνει ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεν δουλεύει θα σας υπολογίσουμε και εσάς ωραία λοιπόν Έληξε η ψηφοφορία. 18 υπέρ, 5 κατά και να μετρήσω και τον συνάδελφο που είναι οπωσδήποτε υπέρ προφανώς. 19 υπέρ, 5 κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπέλετ. Ήταν δύσκολη η δουλειά σας. Madame Βεργιά. Κυρία Εγώ απέχω. Δεν μετρήσατε τις αποχές. Ζητώ συγγνώμη. Δεν, το, δεν βλέπω την οθόνη, λέει η κυρία Πακ πλέον, αλλά υπήρχε μία αποχή. Η επόμενη ψηφοφορία έχει αναβληθεί. Δεν ήταν και τόσο επίγουσα και δεύτερον βεβαίως έπρεπε να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα σε συνεννόηση λοιπόν με την κυρία Καμάεβα αναβλήθηκε και η Επιτροπή Ελευθεριών τόσο ή δεν απέχει τόσο πολύ. Υπάρχει μια ακρόαση την οποία θα πρέπει να περιμένουμε. Οπότε περνάμε τώρα Οπότε περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της Μαρία Μπάντια Ικουτσέτ ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για υποστήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Υπήρχε βεβαίως μια συζήτηση με την Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά καταφέραμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην κυρία Βαδία Ικουτσέτ να ε, ενισχύσει τα σημεία της δικής μας Επιτροπής. Οπότε θα ακούσουμε κάποιες πρώτες σκέψεις και φαντάζομαι πως η κυρία Μπάντια Ικουτσέτ θα μας πει τις ε, σκέψεις της. Παρακαλώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι ήταν σημαντικό που στην Επιτροπή μας ε, θα γνωμοδοτήσουμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Πράγματι πρόκειται για την γνωμοδότηση. Αυτή η καθήλυνα αρμόδια είναι η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Όθηση λοιπόν ε, στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Βάσει του άρθρου 166 λοιπόν της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αναπτύξουμε μια πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση που θα ενισχύει και θα συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών μελών. Η διαδικασία της Κοπενχάγης, η οποία ξεκίνησε το 2002, βοήθησε τα κράτη-μέλη να εξυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και στον τομέα της επαγγελματική κατάρτισης και στα τέλη του 2010 θα γίνει μια συνεδρίαση αξιολόγηση για το πώς έχει η κατάσταση στον τομέα του εξυγχρονισμού της ε, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης και για το πού βρίσκεται η διαδικασία της Κοπενχάγης. Πράγματι θέτει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση για να ε, προωθήσουμε την ανάπτυξη και όπως λέει το κείμενο συγκεκριμένα και βιώσιμη και ευφυή και βέβαια για να το πετύχουμε αυτό είναι πολύ σημαντική η ποιότητα των ανθρώπινων πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού. Και αναφέρεται ότι η αποστολή της μεταγνωτικής εκπαίδευσης είναι διπλή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βοηθήσει να καλυφθούν οι ανάγκες ε, και βραχυπρόθεσμα και μελλοντικά σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και δεύτερον να μειωθεί ο αντίκτυπος της κοινωνικής κρίσης ε, και να βελτιωθεί μελλοντική ένταξη. Και επομένως απαιτούνται διάφορα οι υπουργοί τη ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εκπαίδευση και οι κοινωνικοί εταίροι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσουν στα τέλη Δεκεμβρίου, όπω είπα, τη δρομολόγηση αυτής της διαδικασίας τη Κοπενχάγη. στόχο, λοιπόν αυτή τη ανακοίνωση είναι να προτείνει ουσιαστικά ένα όραμα ε, για το μέλλον στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι ανάγκες που υπάρχουν και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. Πριν σχολιάσω κάποια από τα μέτρα τα οποία προτείνονται, θα ήθελα να επισημάνω ότι θεωρώ ότι η ανακοίνωση αυτή είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε στην Επιτροπή Πολιτισμού ε, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα γιατί σαν υπόψη και ορισμένε από τι δικέ μα εκθέσει. Από την έκθεση που αφορούσε τη βελτίωση τη εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού μέχρι ε, τη ε, διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων, αλλά όχι μόνο για την απόκτηση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, αλλά και για την εφαρμογή του και σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό κλάδο, σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Σε ανακοίνωση λοιπόν, λοιπόν ασχολούνται με θέματα όπως η Ευρώπη 2020 απαιτεί μια στρατηγική για την ενίσχυση της επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης και αυτό το συνδέει με δύο προγράμματα. Το πρόγραμμα των νέων δεξιοτήτων και απασχόλησης και το πρόγραμμα νεολαία σε κίνηση. Νομίζω ότι δεν διαφέρει σε κανένα το γεγονός ότι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα σε ό,τι αφορά ε, την έλλειψη εργασίας ε, είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται πολύ με την εκπαίδευση σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχει ένα ε, διπλό ποσοστό ανεργίας στους νέους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες, με τις υπόλοιπες οικιακές ομάδες. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, ληφθούν μέτρα ιδίω σε σχέση με την νεολαία. Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να απαντήσει ακριβώς, να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Αναφέρονται επίση ορισμένε βασικέ αρμοδιότητε Επιτροπή ε, Πολιτισμού, μόνιμη η διαβίου μάθηση, βασικέ δεξιότητε, νεότητα κτλ. Στο σημείο 2 τη ανακοίνωση η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάγκη να επικαιροποιούνται, να επικαιροποιούνται συνεχώ οι γνώσει. Και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα ε, πρέπει να μπορούν ίσω να συνεχίζουν τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και προγράμματα επαγγελματική εκπαίδευση, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην απόκτηση γνώσεων και επίση και μεγαλύτερη κινητικότητα. Ε, οι εκπαιδευτικοί ε, έχουν ε, ευθύνε, έχουν νέε προκλήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά για την ανάπτυξη τη επαγγελματική εκπαίδευση. Η ανακοίνωση επίση αναφέρει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις βασικές δεξιότητες για την επαγγελματική εκπαίδευση και στους υπόλοιπους ε, κύκλους επιμόρφωσης. Και υπάρχουν εδώ κάποιες αρμοδιότητες που εν γέννη αλλά και πάντοτε σε ορισμένες χώρες είναι πρόβλημα δηλαδή η γνώση ξένων γλωσσών. Νομίζω ότι πολλές φορές στις εκθέσεις μας το τονίζουμε. Τονίζουμε την ανάγκη για την ε, εκμάθηση ξένων γλωσσών. Εκπαίδευση και κατάρτιση λοιπόν προωθούν την κοινωνική ένταξη. Είναι μια πτυχή που λαμβάνεται υπόψη στην ανακοίνωση η ένταξη των ατόμων ε, που έχουν ειδικέ ε, εκπαιδευτικές μαθησιακές ανάγκες, ε, μετανάστες κτλ. ή κάποιοι τομείς που χρειάζονται περισσότερη ειδική βοήθεια. Με την ατυπική μάθηση αλλά και την τυπική μάθηση ε, που λαμβάνεται υπόψη στην ανακοίνωση μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι. Για τους επιχειρηματίες επίσης. Θα πρέπει επίσης να δοθεί σε όλους τους ε, μαθητές στην επαγγελματική εκπαίδευση, ε, κατεύθυνση στον τομέα της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, ε, της επιχειρηματικότητας. Λαμβάνεται επίσης υπόψη διεθνέ επίπεδο η μεγαλύτερη συνεργασία και όχι μόνο με τον ΣΑΛΑ και με τις ε, οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, την UNESCO, Επιστήμη και Πολιτισμός και διάφορα άλλα κέντρα. Και τέλος γίνεται λόγος για το πρόγραμμα Λεωνάρντο Νταβίντσι που είναι το βασικό κοινοτικό εργαλείο υπέρ της επαγγελματική εκπαίδευσης. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την ανακοίνωση, θα την έχετε τη δυνατότητα αυτή και βέβαια θα έχετε σύντομα και το σχέδιο της γνωμοδότησης, το οποίο θα σας παρουσιάσω και εγώ. Με όλα αυτά όμως που σχολίασα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια πληρέστατη ανακοίνωση. Το μόνο που απομένει σε μένα να πω είναι ότι για να μπορέσουν όλα αυτά να εφαρμοστούν, όλες αυτές οι συνταγές, αν θέλετε, τη ανακοίνωση, χρειάζονται πόροι, χρειάζονται επενδύσεις. Και βέβαια, βασικά αυτό είναι απόκειτα στα κράτη-μέλη. Αυτό που με ανησυχεί όμω και θέλω να σα το πω είναι ότι έτσι όπω έχουν τα πράγματα, η κατάσταση, οι προπολογισμοί των περισσότερων κρατών μελών, αυτή η επιστολή που είπε ότι η πρόεδρό μα θα στείλει στου υπουργού ε, παιδεία και πολιτισμού Νομίζω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε ίσως να το ε, έχουμε υπόψη μας, πώς θα βελτιώσουμε την εκπαίδευση των ε, μαθητών μας, αλλά και των ενηλίκων, κάτι που είναι βασικό για να εξέλθουμε από την κρίση, για να έχουμε έναν ε, καλύτερο οικονομικό τομέα, μια καλύτερη οικονομία, πώς θα το πετύχουμε αν δεν συμπεριληφθούν τα σχετικά κονδύλια στο προπολογισμό. Με λίγα λόγια αυτά λοιπόν λέγει η ανακοίνωση. Επίσης κυρία Πρόεδρε νομίζω ότι έχουμε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο την ανακοίνωση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαρία, σας διαβεβαιώ πως ε, έχω λάβει απαντήσεις εντωμεταξύ από τις πρωτεύουσες οι οποίες θα διαβαστούν. Τις έχω δώσει στο Γιούργεν Όλες είναι πολύ φιλικές, όλοι λένε πως έχουμε δίκιο και τώρα δεν ξέρω αν θα τα τηρήσουν όλα αυτά, εν θα το δούμε. Ο μόνος ο οποίος προσπάθησε να τα αρνηθεί όλα αυτά ήταν ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος εξήγησε εκτεταμένα γιατί τα πράγματα δεν μπορούν να είναι αλλιώς. Όλοι οι άλλοι ήταν έτσι κάπως πιο μιχλώδης, έτσι λιγότερο ρητής. Δεν ξέρω, εσύ μπορούμε να πείσουμε τους Γερμανούς. Να δούμε. Ο κύριος Ντελγάδο είναι εδώ από την Κομισιόν. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία, κυρία Πρόεδρε. κυρία Μπαντία αναφέρθηκε στα πιο βασικά σημεία θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι δέκα χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση το 2001 στην Bruges και οι Υπουργοί Παιδείας, οι Υπουργοί που είναι υπεύθυνοι για την ε, επαγγελματική κατάρταση και επιμόρφωση θα επανέλθουν στην Μπρίζ για να κάνουν μια αναθεώρηση, αν θέλετε, των ε, στόχων στα πλαίσια του 2020. Ε, η Κομισιόν θεωρεί την στρατηγική, επανευλα, επανεξετάζει μάλλον την στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη και τους στόχους του προγράμματος του 2020. Θα ήθελα να τονίσω ότι για μας η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση είναι, αποτελεί μια πρόκληση. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Καταρχάς σε σχέση με την κατάσταση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Περισσότεροι άνθρωποι μεγάλη ηλικία θα παραμένουν στην αγορά. Άρα αυτά τα άτομα πρέπει να επανακαταρτιστούν. Και πώς θα γίνει αυτό? με την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση μέσα στα πλαίσια της ε, οικονομικής κρίσης, ε, η ανεργία ανεβαίνει ε, και αν δεν υπάρχει μια επανεκπαίδευση δεν είναι εύκολο τα άτομα να επανέλθουν στην αγορά και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και από την κρίση. Η δεύτερη τάση είναι ο... Είναι ε, οι νέοι μπαίνουν στην αγορά και αυτά τα άτομα και οι νέοι πρέπει να ε, καταρτιστούν. Έχουμε τα στοιχεία του ΣΕΝΤΕΦΟΠ για το 2020 και λέει ότι το 2020 το 50% του πληθυσμού θα έχει μέσης ποιότητας προσόντα. 15% ε, χαμηλά προσόντα και 30% θα είναι εξειδικευμένοι. Άρα θα, η ανάγκη για επιμόρφωση θα είναι κυρίαρχη στην αγορά. Είναι καλό να έχουμε άτομα μορφωμένα από τα πανεπιστήμια κτλ. Όμως τις δουλειές δεν θα τις αποκτήσουν από τα διπλώματα, από τα πτυχία του Πανεπιστημίου, θα τα αποκτήσουν, τη δουλειά θα την εξασφαλίσουν από τα διπλώματα μιας σχολής επαγγελματικής θα πρέπει να καλύψουμε τους τέσσερις πυλώνες ε, της ε, ανακοίνωσης ε, για την εκπαίδευση το 2020, να δούμε ποιος είναι ο βασικός ρόλος της επαγγελματικής κατάρτισης όσον αφορά την διαβίου εκπαίδευση και την κινητικότητα. τα ποσοστά που έχουμε είναι πολύ ε, χαμηλά σε σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση. Η κινητικότητα αποτελεί ένα προνόμιο, νομίζω, για τους, ε, ένα πλεονέκτημα μάλλον για τους εργαζόμενους και καλό είναι θα είναι αυτό να το αποκτήσουν. Καταρχάς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ποιότητα βέβαια, αλλά και να υπάρχει διαπερατότητα ανάμεσα στους διάφορους τομείς. Κάποιος ο οποίος βγάζει μια σχολή επαγγελματική, μετά δεν μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο και αυτό ε, αποτελεί ένα αντικίνητρο και για αυτόν και για την οικογένειά του. Γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν να εφαρμόσουν ένα διαπερατό, αν θέλετε, σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει χαμηλή ποιότητα, αλλά να υπάρχει καλή ποιότητα και δυνατότητα να περνάνε από το ένα σύστημα στο άλλο. Το δεύτερο, δεύτερος πυλώνας είναι η ισότητα. Και αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την εγκατάλειψη σχολείου σε μικρή ηλικία. Όμως, θα πρέπει να βελτιώσουμε και την εικόνα των παιδιών που φεύγουν από τα σχολεία. Θα πρέπει να μπορέσουμε να τους επιτρέψουμε να περάσουν και στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης. Τρίτος πυλώνας δημιουργία και καινοτομία. Θα πρέπει να έχουμε πιο δημιουργική διδασκαλία, πιο δημιουργική εκμάθηση και θα πρέπει να προωθήσουμε, αν θέλετε, και τα επιχειρηματικά προσόντα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις και χρειάζεται να αποκτήσουν επιχειρηματικά προσόντα. Τώρα, ε, θα λάβουμε υπόψη μας ε, τις ιδέες σας και ελπίζουμε ότι τα επόμενα, για τα επόμενα 10 χρόνια η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση θα παίξει ένα πιο αποτελεσματικό ρόλο στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού τοπίου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω πως ε, το, την Παρασκευή ήμουν ε, στην Κοπενχάγη και σας ε, εκπροσώπησα στο 10 επέτειο του Γκρουντβίχτου του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων και διαπίστωσα στη συζήτηση εκεί με τους εθνικούς εκπροσώπους πως χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μία καλύτερη δικτύωση μεταξύ Λεωνάρντο και Γκρούντβιχ γιατί η εκπαίδευση των ενηλίκων βρίσκεται και στα δύο αυτά προγράμματα, και στον Grundwig και στο Λεονάρντο. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ αυτών των δύο προγραμμάτων. Και η Κομισιόν, η οποία ήταν επίσης παρούσα, μου υποσχέθηκε πως το νέο πρόγραμμα διαβίου μάθησης θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες σύνδεσης. Αλλιώς ε, το πρόγραμμα Grundwich δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί πολλές δυνατότητες γιατί είναι πρόγραμμα όπως λέμε επαγγελματικής κατάρτισης αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλες πτυχές. Οπότε παρακαλώ την συνάδελφο τη Μαρία να σκεφτεί πώς θα υπάρξει και μία συνεισφορά στο νέο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε πλέον έτσι με παροπίδες. Π.χ. στην νεολαία σε κίνηση υπάρχει μια ορμή που λέει πως όλα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Γιατί να μην λέμε και ενήλικες σε κίνηση και να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα διάφορα προγράμματα μεταξύ τους. Εάν σκέφτεστε κι εσείς ε, ανάλογα νομίζω θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη νέα γενιά του προγράμματος αυτού διαβίου κατάρτισης. Ο κύριος Μπόρης λοιπόν το λόγο. Ε, dziękuję bardzo za, za ten komunikat. Ε, ja miałem okazję zajmować się między innymi szkolnictwem zawodowym w 3 milionowym με την επαγγελματική κατάρτιση σε μια περιοχή με 3 εκατομμύρια ανθρώπου οπότε έχω άμεση γνώση. Η έκθεση για την Ευρώπη 2020 είναι κάπω θλιβερή γιατί διαβάζουμε εκεί πέρα πω ένα τρίτο των ανθρώπων στην αγορά εργασία δεν έχουν επαγγελματικέ δεξιότητε. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια θεωρώ πως πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως ε, ισχύει αυτό το οποίο είπατε, πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το Λεωνάρντο Νταβίντσι, το Γκρούντβιχ, αλλά θέλω εδώ πέρα να επισημάνω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ ισχυρό δημοσιονομικό εργαλείο που είναι αφιερωμένο στην διαβίω, κατάρτιση και εκπαίδευση. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και νομίζω πως πρέπει να το τονίσουμε αυτό στην έκθεση. Η ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και σήμερα πρέπει να συζητήσουμε το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολωνία με 40 εκατομμύρια πληθυσμό έχουμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ για επαγγελματική κατάρτιση. 12, με συγχωρείτε, δισεκατομμύρια ευρώ σε μια χώρα. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε τους ε, τέσσερις αυτούς ε, πυλώνες για το πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, καλύτερα. Εις ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στις χώρες στόχου 1. Μιλάω λοιπόν για ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τη στρατηγική 2020 και κάτι ακόμα. Εγώ είμαι απόφυτος επαγγελματικός. Ένας απόφυτος επαγγελματικής σχολής θα, μπορεί να θα πρέπει να μπορεί να κάνει βέβαια και μία πρακτική εξάσκηση και να έχει μετά την ευκαιρία να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του αυτές ε, στην ε, πράξη και να συνεχίσει την εκπαίδευση του ή ε, στην ανώτατη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι αρκετά ανοιχτή, το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε αρκετή εσωτερική μετανάστευση και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ξένες γλώσσες και η διαδικασία αυτή βεβαίω ακόμα είναι μπροστά μας. Ξέρω πως η Γερμανία, η Αυστρία έχουν ανοίξει την αγορά εργασίας και πρέπει να θυμόμαστε πως αυτό δεν αφορά μόνο όσους έρχονται εκτό Ευρώπης, αλλά είναι ήδη εντό της Ευρώπης. Ευχαριστώ την Μαρία Μπαντία για την έκθεση, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας, όπως είπε και η πρόεδρος Πάκα, Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την Κοπενχάγη και η Επιτροπή μας ε, πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της στο θέμα αυτό, διότι είναι ένα από τα θέματα που, στο οποίο δεν έχουμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Η διαβίου εκπαίδευση και η σχέση της επαγγελματικής κατάρτισης και διαβίου ε, διαβίου κατάρτισης με την ε, επαγγελματική αποκατάσταση δεν ε, υπάρχει. Θα πρέπει δηλαδή να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και όπως είπε η κυρία Μαντία θα πρέπει να κάνουμε κάποιες υπερβάσεις. Καταρχάς και στην χώρα μου υπάρχουν εμπειρίες πολύ πετυχημένες από, την, από το πέρασμα από το σχολείο στα, στην ε, επαγγελματική εκπαίδευση και την επιστροφή. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες πασαρέλες που επιτρέπουν το τελικό αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο θετικό. Και τα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν τι τους γίνεται από τα 15 του στα 18, δηλαδή καταλείπουν το σχολείο ή δεν ξέρουν τι θα κάνουν, μπορούν να πάνε στα επαγγελματικά, στις επαγγελματικά λύκεια αν θέλετε και με, εάν δεν το αλλάξουν γνώμη μπορούν να επιστρέψουν πάλι στο σχολείο και να πάρουν το πτυχίο τους. η Κομισιόν είπε ότι υπάρχει και ένα θέμα εικόνας τη επαγγελματική της επαγγελματικής κατάρτισης, των, ε, ε, των επαγγελματικών ηλικίων. Ε, αυτό μπορεί να ισχύει σε κάποιες χώρες, αλλά νομίζω ότι αυτή την εικόνα θα πρέπει να την αποκαταστήσουμε, διότι αν δούμε τι ζητάνε οι επιχειρήσεις και τι ζητάει η βιομηχανία, αυτό το οποίο ζητάνε είναι προσόντα, προσόντα εξειδικευμένων εργαζομένων. Επομένως, τα συστήματα θα πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και κυρίως ε, σε επίπεδο μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στα σχολεία και στην ε, αγορά. Θα πρέπει επίσης, όπως είπε και η Μαρία Μαντία, να ε, φέρουμε μαζί και να δημιουργήσουμε κάποια δίκτυα, κάποιους συσχετισμούς, δεν ξέρω, καθένας θα βρει τον, τον τρόπο ε, που θα το κάνει, ε, ανάμεσα στα επαγγελματικά ιδρύματα, στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε και την υπόψη μας και τη θέση των γυναικών. Ούτως ή άλλως τα κορίτσια ε, ε, είναι πολύ πιο ομορφωμένα και πολύ έχουν περισσότερα ε, πτυχία κτλ. Όμως στα προσόντα, στα επαγγελματικά προσόντα, στην επαγγελματική εκπαίδευση εκεί υπάρχει, υπάρχει ένα έλλειμμα αν θέλετε γυναικών. Δηλαδή είναι περισσότεροι άντρες από τις γυναίκες σε τέτοιου είδους, ε, σε αυτού εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Την ε, κυβέρνηση της Ουγγαρίας έκανε κάποια βήματα για την ε, αναδιάρθρωση του συστήματος επαγγελματική κατάρτισης όταν προέκυψε ότι δεν ήταν επιτυχημένο το τωρινό σύστημα. Δεν συνέπειπτε η προσφορά με την ζήτηση. Υπάρχουν προβλήματα στο συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και στις επιθυμίες των νέων, στο τι θέλουν να σπουδάσουν και αν αυτό το ζητάει η αγορά. Οι έρευνες, οι προσανατολισμένες προς την αγορά έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν και εδώ πέρα πρέπει και εμείς να εμπλακούμε γιατί πρέπει να αποφευθεί το να εκπαιδεύουμε με ακριβό τρόπο ανθρώπους για επαγγέλματα τα οποία δεν ε, ζητάει η αγορά. Ίσως να μην είναι γενικό το πρόβλημα, αλλά στην Ουγγαρία η επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ θεωρητική και υπάρχει και το ζήτημα της επανεκπαίδευσης και των διδασκόντων οι οποίοι συχνά έχουν απερχιωμένες ε, γνώσεις και πρέπει να αλλάξουν οι τεχνικές ε, και η στρατηγική. Πρέπει λοιπόν να γίνει ίσως μία σύσταση για τις ε, διάσημες αυτές οι διαβόητες βέλτιστες πρακτικές τις οποίες θα πρέπει να μιμηθούμε και καλό θα ήταν να γίνει μια σύσταση στο κείμενο αυτό για τους διδάσκοντες οι οποίοι θα πρέπει επίσης ε, να έχουν μία διαβιοκατάρτιση Δεν αρκεί ένα πτυχίο που πήραν κάποτε και θα πρέπει νομίζω να αναφέρουμε πως ε, αυτό που σας είπα, οι δάσκαλοι, σχολεία να εκπαιδεύονται περαιτέρω και να υπάρχει κινητικότητα όχι μόνο μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των διδασκόντων. Νομίζω και αυτό είναι σημαντικό. Θεωρώ πως ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για εποχιακά επαγγέλματα, εποχιακά επαγγέλματα που αφορούν είτε μία εποχή του χρόνου είτε μία περίοδο ετών. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να έχουν μόνο μία κατάρτιση οι νέοι, αλλά ίσως περισσότερες για να μπορούν να έχουν μία μόνο εποχιακή εργασία, αλλά δύο ίσως να απασχολούνται και κάπου αλλού. Στην Ουγγαρία, λοιπόν, όπως σας έλεγα, κάθε επιχείρηση πληρώνει μια συνεισφορά στο Ταμείο Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα. Γι' αυτό θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες ε, πρακτικού προσανατολισμού της επαγγελματικής κατάρτισης σε ένα διπλό σύστημα έτσι ώστε να μάθουν μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά πράγματα. Thank you, Madam. I will be brief. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Θέλω να τονίσω τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτισης. Η διαδικασία της Κοπενχάγης που είναι ίσως ε, η μεγαλύτερη πιο σημαντική διαδικασία στον τομέα τη εκπαίδευση είναι σημαντική. Νομίζω ότι μπορούμε να συγκρίνουμε τη διαδικασία τη Κοπενχάγη με τη διαδικασία τη Μπολόνια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση νομίζω ότι ως τμήμα της εκπαίδευση θα πρέπει να εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη δεκαετία. Ο σκιώδης εισηγητής προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους μου για το θέμα αυτό, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σήμερα κάνει κάποιες ε, υποθέσεις, παρουσίασε κάποια σενάρια τα οποία είναι πολύ καλά και νομίζω ότι από κοινού μπορούμε να βελτιώσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εντός της προσεχούς ε, δεκαετίας. και να την εντάξουμε στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις που πηγαίνουν προ την κατεύθυνση της Ουγγαρέζας ε, συναδέλφου. Γνωρίζουμε όλοι πως δεν μπορούν οι πάντες να γίνουν πανεπιστημιακοί και δεν πρέπει. Κάποιος πρέπει να φτιάξει τα πλακάκια, τη θέρμανση, τη στέγη, Χρειαζόμαστε λοιπόν και χειρόνακτες οι οποίοι θα είναι σωστά εκπαιδευμένοι για να μπορούν να σταθούν στην εσωτερική αγορά και γι' αυτό χρειάζονται μια ξένη γλώσσα. Εγώ προέρχομαι από μια μεθοριακή περιοχή, όπως και πολλοί από σας. Είναι αδύνατον οι νέοι άνθρωποι να μην μιλάνε την γλώσσα των γειτόνων μας για να μπορούν να πάνε και να κάνουν προσφορά ή να λάβουν μέρος σε ένα διαγωνισμό στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο. Γι' αυτό συμφωνώ με τη Μαρία. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, το θέμα ξένες γλώσσες στην επαγγελματική κατάρταση έχει μεγάλη σημασία, αλλά όχι όπως ε, διδάσκεται ή διδάσκονταν παλιά στο σχολείο, αλλά να συνδεθεί με την πράξη. Ο νέος ο οποίος θέλει να γίνει υδραυλικός ή φλακάς πρέπει να ξέρει τις εκφράσεις της δουλειάς. Χρειαζόμαστε δηλαδή επικέντρωση στις ξένες γλώσσες, ειδικά στις μεθοριακές περιοχές της γλώσσας της γειτονικής χώρας και δεύτερον, καλύτερη κατάρτιση των διδασκόντων. Υπόθηκε πολλές φορές. Το είπα πως ε, χρειάζεται και έχουμε ένα νέο κομμάτι στο κομμένιους που λέγεται κομμένιους για τους δασκάλους που θα συμπεριλάβει τους δασκάλους. Και νομίζω εκεί πέρα θα έχουμε ακριβώς μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, δηλαδή στο θέμα των γλωσσών. Σας παρακαλώ λοιπόν να το σκεφτείτε αυτό και να συμπεριλάβετε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Εάν όχι, εντάξει, θα καταθέσουμε τροπολογίε, αλλά νομίζω πω ε, πίστηκε η Μαρία πω είναι σημαντικό αυτό. Εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, η Μαρία θέλει να πει τίποτα άλλο. Είμαι εδώ πέρα. Θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, έτσι πιστεύω τουλάχιστον, αυτό το θέμα. Συμμερίζομαι όλες τις ε, σκέψεις ε, και ανησυχίες σας και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ουσιαστικά τα ε, είπατε όλα, αλλά πολύ σημαντικό ήταν αυτό που είπατε, να δώσουμε ένα μεγαλύτερο γόητρο, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη αξία στην επαγγελματική εκπαίδευση. Έχουμε δει τι γίνεται στι χώρε. πώς αναπτύσσουν αυτά τα προγράμματα. Έχουμε δει τι γίνεται στι οικογένειε. Όταν ε, ο γιος ή η κόρη λέει ότι δεν θέλει να πάει στην, ε, στο πανεπιστήμιο, αλλά ε, θέλει να κάνει επαγγελματική σχολή, νομίζουμε ότι είναι δευτέρα ή τρίτη κατηγορία οι σπουδέ που θέλει να κάνει το παιδί μα. Γιατί λοιπόν γίνονται όλα αυτά. Γιατί δεν θεωρείται καλή εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Άρα αν καταφέρουμε να αλλάξουμε την οτροπία, ότι δηλαδή το να μάθει κανείς ε, το επάγγελμά του δεν σημαίνει ότι κάνει κατώτερες σπουδές, αλλά ότι ουσιαστικά οι σπουδές του είναι του ίδιου επίπεδου, όπως ε, αν πήγαινε στο πανεπιστήμιο. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, δεν αλλάζει τίποτα. Πώς θα το πετύχουμε. Θα το πετύχουμε αν έχουμε καταρτισμένους εκπαιδευτικούς ε, που παρέχουν ποιοτική διδασκαλία και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα μετάβαση, οι γέφυρε, όπω είπαμε. Δηλαδή, να ξεκινήσει ο μαθητή από την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά αυτό να μην του κλείσει την πόρτα για το Πανεπιστήμιο, αν τον ενδιαφέρει στο μέλλον. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ε, γιατί πολλές φορές ο κόσμος ε, λειτουργεί ε, με τα συναισθήματα, αν είναι ικανοποιημένος με αυτό που κάνει. Αν δεν αλλάξει αυτή η ιδέα ότι η επαγγελματική εκπαίδευση είναι εκπαίδευση δεύτερης κατηγορίας, δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Όλα όσα σχολιάσατε αγαπητοί συνάδελφοι με βρίσκουν απόλυτο σύμφωνοι. Ίσως το πρόβλημα θα είναι ότι όπως γνωρίζετε η γνωμοδότηση ουσιαστικά είναι μια σελίδα κείμενο. Άρα ε, το θέμα είναι να αποφασίσω τι θα συμπεριλάβω ως προτεραιότητα σε αυτή τη μία σελίδα αλλά νομίζω ότι όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι και οι συνάδελφοι στην Επιτροπή εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε καλή δουλειά. Και φυσικά δεν τελειώνει εδώ η προσπάθεια, είναι ένα θέμα που θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και αν στα τέλη της χρονιάς έχουμε και την αναθεώρηση της διαδικασίας της Κόπενχάγης, θα συνεχίσουμε τη σχετική συζήτηση. Ένα σχόλιο, αν με επιτρέπετε, δεν ξέρω ποιο το είπε, νομίζω ο Σκιώδη, ε, εισηγητή, ε, μίλησε για τη σύγκριση μεταξύ τη διαδικασία τη Μπολόνια και τη διαδικασία τη Κοπενχάγη. Νομίζω ότι αν κάνουμε αυτή τη σύγκριση και αν μιλήσουμε για ανάγκη εναρμόνισης ε, σε, ως έναν βαθμό συμφωνώ. Αν όμως ε, το συγκρίνουμε με την κοινωνική αντίληψη της μίας και της άλλης διαδικασίας, νομίζω ότι είναι εντελώ διαφορετικά τα πράγματα. Η διαδικασία της Μπολόνια αμφισβητήθηκε ιδιαίτερα σε πολλές χώρες της Ένωσης. Και αυτό διότι ο στόχος ουσιαστικά ήταν να εκφράσουμε τις απόψεις και να αξιολογήσουμε κάποιες ακαδημαϊκές, ε, πανεπιστημιακές ε, σπουδές που είναι top, που είναι η κορυφή. Εμείς είμαστε ανώτεροι και πώς θα κάνουμε άλλοι, πώς θα συγκριθούμε με κάποιον. Η μικρή αδερφή ή ο φτωχός συγγενής αν θέλετε, η επαγγελματική εκπαίδευση δηλαδή, χαίρεται ιδιαίτερα άμα την προσέξει κανείς ε, και της δώσει σημασία. Άρα το να ε, γίνει εναρμόνιση σε έναν βαθμό, ναι, μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση. Αλλά σε ό,τι αφορά την κοινωνική αντιμετώπιση, νομίζω ότι αντίθετα από την ανώτερη εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση θα χαρεί αν τη δίνουμε βοηθεία. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εμεί δεν είχαμε εμπλακεί στην Πολώνια, στη διαδικασία τη Πολώνια. και τώρα είναι αλλιώ τα πράγματα και όπω λέ, πρέπει να φροντίσουμε το αποπέδι αυτό να το φροντίσουμε κάπως περισσότερο. Και βλέπουμε στους στόχους στρατηγικής 2020 πως δεν αναφέρεται τίποτα από αυτού. Μιλάμε για όσους ε, φεύγουν από τα σχολεία νωρίτερα, να μειωθούν αυτοί και να ανεβούν κατά 5% από αυτή πανεπιστημίου. Και πού είναι αυτό το οποίο τελικά αποτελεί την καθημερινότητα δεν αναφέρεται πουθενά παρά το ότι μιλάμε παντού για απασχόληση, αλλά αυτό το οποίο θα μπορούσε να φροντίσει το θέμα αυτό και αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να απασχοληθούν δεν αναφέρονται πουθενά. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε το μέσα αυτός να έρθει στο προσκήνιο. Και εδώ πέρα μπορώ να σε καθυσυχάσω, είμαστε σύμφωνα Είμαστε σε μια διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 50, είμαστε δηλαδή μια συνδεδεμένη επιτροπή, μπορείς να γράψεις πάνω από μια σελίδα. Άρα, αν θες να εισαι συντομη σύντομη, γράψε μια-δύο σελίδες. Αλλά νομίζω πως πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το οποίο είναι σημαντικό, όχι σε αυτό το οποίο θα κάνει ούτως ή άλλως η κοινωνική επιτροπή. Οπότε νομίζω πως έχουμε περισσότερες δυνατότητες εδώ πέρα υπ' αυτό το καθεστώς. Οπότε ευχαριστώ Μαρία και καλή επιτυχία. Περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε μία γνωμοδότηση για το θέμα «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» από την Επιτροπή ε, αλλά βεβαίω έχει μία πτυχή πολιτισμού που είναι σαφής, οπότε κάνουμε μία γνωμοδότηση και η κυρία Ράνερ θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ντόρις, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα προσφέρεται ακριβώς όπως έδειξε και η συζήτηση για να τοποθετηθούμε εμείς γιατί όπως θα πω και εδώ πέρα το θέμα αφορά την κατάρτιση πάρα πολλών ανθρώπων που δεν ε, έχουν κάποιο πανεπιστημιακό πτυχίο αλλά κάποια άλλη εκπαίδευση. Όπως ε, είπες ε, εδώ πέρα η κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Μεταφορών αλλά και εμείς συμμετέχουμε στην γνωμοδότηση. Αν δείτε λοιπόν την ανακοίνωση της Κομισιόν που είναι πολύ λεπτομερής, βλέπουμε ακριβώς το πρόβλημα εδώ πέρα του θέματος. Ο τουρισμός δίνει ε, δυνατότητες βεβαίως ε, απασχόλησης μερικής ε, μπορεί να είναι περιφερειακός, εθνικός, πολιτιστικός. Προσπάθησα λοιπόν να επικεντρωθώ εγώ στον δικό μας τον τομέα αρμοδιότητας γιατί θεωρώ πως αυτό είναι το σωστό. Αλλιώς θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό. Αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που έχουμε εδώ πέρα και να προσπαθήσουμε να βρούμε καινοτόμε λύσεις για να παραμείνουμε πρωτοπόροι από τη Λισαβόνα και μετά έχουμε κάποιες νέες αρμοδιότητες. Ο τουρισμός λοιπόν πάρα πολύ σημαντικός και βεβαίως, όπως λέμε, η κληρονομιά είναι ένα θέμα, η χρήση της είναι κάτι άλλο. Μιλάμε για 1,8 εκατομμύρια ε, επιχειρήσεις πάνω από το 5% του ΑΕΠ ε, άμεσα και των θέσεων εργασίας και μιλάμε για 10% ε, των θέσεων εργασίας ε, πραγματικά και αποτελεί έναν κινητήρα οικονομικής ανάπτυξης, κάτι το οποίο συνδέει τα κράτη-μέλη, γιατί βεβαίως όποιος εκπαιδεύεται στον τουρισμό θα πάει στο εξωτερικό, πρέπει να μάθει γλώσσες ε, και να πάει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και εκτός Ευρώπης ε, και το ξέρω αυτό πάρα πολύ καλά γιατί ξέρετε πως η Αυστρία έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά τον τουρισμό, η Αυστρία ζει από τον τουρισμό, αν θέλετε, και χωρίς αυτόν θα είχαμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αλλά ο τουρισμός βεβαίως ε, το δικό μας το θέμα είναι ο πολιτισμός. Ο τουρισμός λοιπόν περιλαμβάνει τον πολιτισμό και στην πτυχή της εκπαίδευσης ε, και στην πολιτισμική κληρονομιά και στην προστασία της ε, φύσης ε, και στα ΜΜΕ βεβαίως και τον αθλητισμό και έχει και πτυχές νεολαίας. Προσπάθησα να αναφέρω κάποιες κατηγορίες τουρισμού και βεβαίως δεν νομίζω να μπορούμε να απομονώσουμε τον πολιτισμό από αυτό το θέμα. Σκεφτείτε τον πολιτισμικό τουρισμό, τι γίνεται με τα μνημεία που πάει ο κόσμος, αλλά και το θερινό, χειμερινό τουρισμό, τα σπα και τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης που έχουμε αναπτύξει και εμείς βεβαίως και επίσης, ναι, ναι προσπαθώ και η Ευρωπαϊκή Σφραγίδα Πολιτισμικών Αγαθών δεν ξέρω τώρα φοβάμαι πως υπάρχει ένας πληθωρισμός εδώ πέρα ευρωπαϊκών σφραγίδων και σημάτων αλλά εν πάση περιπτώσει χρειαζόμαστε λοιπόν κατά τάξη πρέπει να βοηθήσουμε και τον καταναλωτή αλλά δεν είναι δυνατόν βεβαίως ε, να μην παίξει κάποιο ρόλο εδώ πέρα και η αγορά. Η Κομισιόν έχει προτείνει πάρα πολλές δράσεις ε, και μια σφραγίδα βεβαίως ε, και ποιοτική και μια χάρτα για τον τουρισμό. Θεωρώ λοιπόν πως πρώτα απ' όλα να δούμε τις ανάγκες τις ευαισθησίες και τις προτιμήσεις των τουρισμών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με πιλωτικά έργα τα οποία βεβαίως κάνουν εν μέρη και τα κράτη-μέλη και οπωσδήποτε απαιτείται να ανταλλάσσουν πληροφορίες στα κράτη-μέλη πολύ περισσότερο όλα αυτά θα βοηθήσουν να αποκτήσει ουσία αυτή η γνωμοδότηση. Στη δράση υπαριθμών 3, παραδείγματο χάρη, αναφέρεται η σύσταση ενός δικτύου πληροφορικής και επικοινωνίας για τον τουρισμό μια τέτοια πλατφόρμα. Εντάξει, επί της αρχής καλό είναι, αλλά τι μορφή θα έχει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να μας απασχολήσει παραδείγματος χάρη για 20 χρόνια. Μετά στην δράση 90 μιλά για ένα ευρωπαϊκό πόρταλ τουρισμού που θα λέγεται visiteurope.com. Το έχετε ακούσει ή όχι ποτέ σας. Ωραίο ακούγεται. Οπότε θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Και να δούμε βέβαια τι θα περιέχεται εκεί πέρα στο visiteurope.com. Όπως σας είπα είναι πολλά υποσχόμενα αλλά άδειο μέχρι στιγμή το όνομα, η διεύθυνση αυτή. Δράση 11. Αναφέρονται τα προγράμματα NEC Tour και Eden που θα πρέπει να στηρίξουν τη δικτύωση. Άγνωστα για αυτά, τα έχετε ακούσει ποτέ, Νεκ και Όχι. Κανείς. Λοιπόν, αυτές οι πρωτοβουλίες είναι κάπως προβληματικές, ε, γιατί τι γίνεται, έτσι, είναι εδώ και εκεί μια σταγόνα στον ωκεανό. Και θα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν, δεν ξέρω, λίγη περισσότερη χρηματοδότηση, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερη συνέργεια μεταξύ των περιφερειών, των περιφερειακών δράσεων, όπως αναφέρεται και στη δράση υπαριθμών 20, που μιλάμε εδώ πέρα παραδείγματο χάρη για εκδηλώσεις, ε, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, την ε, έκθεση του Βερολίνου για τον τουρισμό, και πρέπει εκεί πέρα να προωθεί περισσότερο ευρωπαϊκό τουρισμό. Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω να υπάρξει και να ενισχυθεί τουριστική εκπαίδευση. Αυτό αφορά πρώτα απ' όλα τις ξένες γλώσσες, αλλά και εκπαίδευση στην ίδια τη χώρα. Στην Αυστρία έχουμε πολλές γνωστές τουριστικές σχολές, αλλά δεν υπάρχουν ανταλλαγές πρέπει να ενισχυθούν πάρα πολύ. Πολλές φορέ έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις εδώ πέρα και διαφορετικές εμπειρίες. Εμείς στην Αυστρία, παραδείγματο χάρη, έχουμε το θετικό. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από την Ανατολή. Οπότε κάποιος τουλάχιστον σε ένα ξενοδοχείο πρέπει να ξέρει ρωσικά. Αλλιώς βέβαια και τόσο θετική εμπειρία, οπότε πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ανταλλαγές. Έτσι, πληροφοριακά, το 2009 εμείς είχαμε πάνω από 13.000, δηλαδή πάνω από 12% όλων των μαθητευομένων ήταν στον τομέα του τουρισμού. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα και το άλλο θέμα που έχουμε αναφέρει, ο εθελοντισμός. Ξέρουμε πως είναι κάτι το σημαντικό για τους νέους και είναι απολύτως απαραίτητο για να πάνε στο εξωτερικό, αλλά γνωρίζουμε πως όλο και συχνότερο, συχνότερα συχνά χρησιμοποιεί το εθελοντισμό για, να πληρω... για να μην πληρώσουν τους νέους ανθρώπους για δουλειά που θα έπρεπε να πληρωθούν. Οπότε νομίζω και αυτό εδώ πέρα κολλάει στην εκπαίδευση του τουρισμού. Μου φαίνεται λοιπόν πως είναι απολύτως απαραίτητο. Κατόπιν το αγαπημένο μου θέμα, το οποίο ε, έχω αναφερθεί πολλές φορές, ε, το οποίο βεβαίως αφορά τα των ε, διακοπών και το πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτά τα τεράστια μποτιλιαρίσματα στην Αυστρία πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με το πότε παίρνει ο κόσμος άδεια. Γιατί αυτό είναι σημαντικό βεβαίως και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις και για όλους. Να δούμε επίσης και το συνεδριακό τουρισμό γιατί βεβαίως εδώ πέρα δημιουργεί προβλήματα οικονομική κρίση, γιατί οι συνέδρια διοργανώνται όταν υπάρχει βεβαίως κάποια ευχέρεια και έχουμε και το λεγόμενο κοινωνικό τουρισμό, δεν ξέρω στα γερμανικά μου βγείτε κάπως περίεργο, αλλά έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι ας πούμε πάνω από 50 ετών και είναι συνταξιούχοι και εάν δεν έχουν επαρκές εισόδημα θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα και το χρόνο να καλύψουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα θέμα νομίζω το οποίο αφορά την Επιτροπή μας και θα πρέπει να το δούμε. Τα υπόλοιπα λοιπόν προγράμματα εκπαίδευσης θεωρούν πως αφορούν την νεολαία και να επικοινωνήσουν οι νέοι. Τι θα γίνει με τους ηλικιωμένου που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε άλλες χώρες και να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες σκέψεις που έκανα στο θέμα αυτό. Όπως σας είπα υπάρχουν εκατοντάδες ακόμα. Νομίζω πως το βασικό εδώ πέρα σε αυτή την γνωμοδότηση θα είναι να δώσουμε κάποια ουσία, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες θα ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και αναμένω τη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Χέλα. Ναι, κοίτα, ε, αυτό τώρα με το να παίρνουν διαφορετικό χρόνο διακοπέ ο καθένα δεν, δε θα αλλάξει το καλοκαίρι. Όλοι το καλοκαίρι θέλουν να πάνε διακοπέ, δεν μπορεί να επιμηκυνθεί. Τι να κάνουμε. Ε, δηλαδή να το ζητήσουμε, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά κάτι το οποίο ε, θα έπρεπε να αναφέρεις νομίζω είναι το εξής. Δεν χρειάζεται να εφευρίσκουμε πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Κομισιόν. Υπάρχει κάποιος υπάλληλο θέλει να κάνει κάτι και λέει «Α, θα κάνω κάτι καινούριο». Γιατί να εφεύρουμε συνεχώς κάτι καινούριο. Έχουμε τα πολιτιστικά δρομολόγια, μία εφεύρεση του Συμβουλίου της Ευρώπης και εγώ τυχαίνει να γνωρίζω πως ε, το προσκύνημα αυτό στο Σαντιάγκο Κομποστέλα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω έναν δημοσιογράφο που έφυγε ένα χρόνο και ακολούθησε την διαδρομή αυτή. Και πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Υπάρχουν αυτοί οι δρόμοι, αυτά τα δρομολόγια που δεν τα ξέρουμε ίσως. Γι' αυτό θα αναφέρω κι εγώ κάτι που βρίσκεται στις νέες χώρες, στη Ρουμανία. Οι εκκλησίες εκεί πέρα στα χωριά, χωριά τα οποία είναι μια εκκλησία και γύρω γύρω τα σπιτάκια μέσα σε ένα τείχος, δηλαδή έτσι οχυρωμένα χωριά με μια εκκλησία στο κέντρο για να προστατευτούν από τον εχθρό και υπάρχει αν θέλετε μια διαδρομή που πηγαίνει ε, από χωριό σε χωριό. Θα έπρεπε αυτό να σε αυτό το πόρταλ στο visiteurope.com και είναι κάτι το οποίο δεν κοστίζει πολύ αλλά μπορούμε να δώσουμε έτσι κάποια δημοσιότητα. Βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουμε και τα χωριά αυτά να ε, δικτυωθούν. Εγώ επισκέφθηκα τρία τέτοια χωριά γύρω από το Σιμπίου και μπορώ να σου πω πως αξίζει τον κόπο. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε ε, να κάνουμε. Οπότε, Χέλα, εάν εστιαστείς λοιπόν σε πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό, νομίζω πως μπορείς να επιτύχεις κάτι στην Επιτροπή Μεταφορών. Ο Μπόρις τώρα, παρακαλώ. Pierwszy wniosek, myślę, że w ogóle turystyka powinna E, το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο θα πρέπει να ε, καταλήξουμε είναι ότι εμείς είμαστε η καλύτερη επιτροπή, η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και όχι η επιτροπή μεταφορών. Αλλά τέλος πάντων αυτό θα το ρυθμίσουμε στο μέλλον. Επί του παρόντος η Ευρώπη δεν προωθεί την ε, ε, την, Ήπειρό μας σαν Ευρώπη, αυτή καθεαυτή. Κάθε χώρα βέβαια προωθεί τον τουρισμό της, όμως θα πρέπει να προωθούμε και τον ε, ευρωπαϊκό τουρισμό και εκτός Ευρώπης, δηλαδή να ε, προσελκύουμε τουρίστες από άλλες υπήρους, όμως θα πρέπει να ευνοήσουμε και τους ε, Ευρωπαίους τουρίστες, δηλαδή οι Ευρωπαίοι να ταξιδεύουν στην Ευρώπη χρησιμοποιήσουμε το, αν δημιουργήσουμε αυτό το πόρταλ ή αυτό το site για την, για την Ευρώπη, ε, θα πρέπει να αναφέρουμε εκεί και τα διάφορα αξιοθέατα. Επίσης, ε, υπάρχει και το θέμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ε, θα πρέπει να υπάρχει και ένα link και μια, ένα, να γίνει και μια, ένα συσχετισμός ανάμεσα σε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και, στην, ε, και στον τουρισμό. Επίσης έχουμε και ένα σωρό αξιοθέατα τα οποία χρειάζονται βοήθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και η πολιτική συνοχής ε, η οποία ακόμα εφαρμόζεται ιδίως στις περιοχές του Νότου έτσι ώστε ναι μεν υπάρχουν κάποια αξιοθέατα τα οποία ήδη την χάνουν υποστήριξης, υπάρχουν και άλλα όμως τα οποία θα πρέπει μέσω της πολιτικής συνοχής η οποία εφαρμόζεται να βοηθηθούν. Υπάρχει και μια εξωτερική υπηρεσία, αν θέλετε, που λειτουργεί λίγο πολύ σαν πρεσβευτής της Ευρώπης θα πρέπει ε, να όταν λέω εξωτερικές υπηρεσίες εννοώ τις πρεσβείες μας, ε, τα προξενία μας ε, και αυτοί θα πρέπει να προωθούν την Ευρώπη σαν τουριστικό προορισμό. Επίσης, αυτά τα ευρωπαϊκά μονοπάτια, ας πούμε, του Σαντιάγκο, τον Κοποστέλα. Επίσης, τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό μονοπάτι, το μονοπάτι των ταγμάτων. Υπάρχουν και διάφορα άλλα μονοπάτια, τέλος πάντων, σε διάφορους τομείς. Αυτά τα μονοπάτια διασχίζουν πολλές χώρες. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε και τουρίστες και εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα νομίζω και μια προοπτική. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλού να Παρακαλώ να είστε Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει τα θέματα του τουρισμού να τα αναλάβουμε εμείς. Γιατί νομίζω μας αφορά πλήρως, γρήγορα να τα πω όλα. Εμεί, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό, αυτό το θέμα των πολιτιστικών διαδρομών να τα προωθήσουμε ιδιαίτερα διότι προωθούμε μια ιδέα του τουρισμού, του πολιτιστικού, του ευρωπαϊκού τουρισμού, πολιτιστικού. Και ε, ζώντας αυτή την οικονομική κρίση την οποία ζούμε τώρα, ο πολιτιστικός τουρισμός έχει αυξηθεί και τα κράτη έχουν αρκετά σημαντικά έσοδα από τον τουρισμό αυτό και άρα θα πρέπει και η προσφορά και η ζήτηση να ευθυγραμμιστούν. Επίσης, σε σχέση με αυτά που είπε και συνάδελφος προηγουμένως, η Μαρία Μπαντία, το θέμα της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό και, και στον τουρισμό, γιατί πολύ λίγα πανεπιστήμια στην Ευρώπη έχουν μαθήματα που αφορούν τον τουρισμό, έχουν τουριστικές σπουδές. Αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, διότι ε, προωθώντας και τις τουριστικές σπουδές αυξάνεται και η ποιότητα των υπηρεσιών, άρα μπορεί να αυξηθεί και η τουριστική κίνηση. Επίσης υπάρχει και ο κοινωνικός τουρισμός, όπως είπε η κυρία Ράνερ, και ο αλληλέγγυος τουρισμός, όχι δηλαδή μόνο ο τουρισμός ο οποίος απευθύνεται στους ηλικιωμένους ή στα άτομα τα οποία δεν έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, αλλά ε, και όλα τα, αλλά και ο τουρισμός ο οποίος απευθύνεται ε, και στα άτομα γενικότερα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη πόσες παραλίες έχουν ε, δυνατότητες πρόσβασης για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να μπορούμε να παρέμβουμε έτσι ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές δυνατότητες πρόσβασης λαμβάνοντας υπόψη ε, όλη τη δουλειά που κάνουμε και για, το, για την ευρωπαϊκή κληρονομιά, την πολιτιστική κληρονομιά Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να το δουλέψουμε το θέμα, έστω και αν η ανακοίνωση της Κομισιόν μου φαίνεται αρκετά λεπτομερής, αρκετά σαφής, δίνει προς προσανατολισμούς, για να μην πω ότι και ε, κάνει και κάποιες επαναστατικές τομές στον τομέα αυτό. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Χέλα τις πολλές πτυχές ε, που ανέδειξε του τουρισμού και τη σημασία που έχει για τον πολιτισμό στην Ευρώπη, αλλά και αντιστρόφως. Θεωρώ όμως πως σημαντικό είναι να συγκεντρωθούμε σε πράγματα που ξέρουμε. Η ποικιλία που υπάρχει, π.χ. θα μπορούσε να αφορά και βιβλία και τέτοια. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η το πώς θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και δυνατότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν διάφορα site ε, που έχουν ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορα έργα ε, τουρισμού ή πολιτισμού και ποιος ξέρει τι υπάρχει πραγματικά εκεί έξω. Οπότε σημαντικό είναι ένα πόρταλο όπως αυτό το οποίο αναφέρατε για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες και πληροφορίες από περιφέρειες για οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς για ποδηλατικό τουρισμό, για ποτάμια. Για το σημαντικό να τα βρει κανείς όλα αυτά, μια σημαντική πτυχή ενίσχυσης ε, του τουρισμού. Για να μπουν όλα αυτά σε ένα πόρταλ και να βγουν προς τα έξω και όσοι βεβαίως ενδιαφέρονται να επισκεφθούν ε, διάφορα πολιτιστικά μνημεία στην Ευρώπη να το βρίσκουν εύκολα. Και οτιδήποτε βέβαιος αφορά τον πολιτισμό και την κληρονομιά νομίζω είναι κάτι το οποίο μας αφορά και δεν πρέπει να το αφήσουμε μόνο στα κράτη-μέλη. Kilka rzeczy, o których Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά αξίζει να υποστηρίξουμε τον τουρισμό και δι για τους ηλικιωμένους, για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τον εσωτερικό τουρισμό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πρέπει να το στηρίξουμε. Θα ήθελα μόνο μία κριτική να ασκήσω. θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε ε, σε συγκεκριμένα ζητήματα, παραδείγματος χάρη υποδομές για τα άτομα με αναπηρία ή μήπως γενικότερα ε, πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων. Η πρόθεση του ευρωπαϊκού τουρισμού, του πανευρωπαϊκού τουρισμού, θα έλεγα ότι είναι ένα παράδειγμα υπερρύθμισης, ένα ακόμα από τα πάμπολα παραδείγματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο λοιπόν, απόλυτα απαραίτητο αυτό. Να έχουμε έναν ακόμα ευρύ τομέα ε, τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί και άλλα όχι τόσο. Νομίζω ότι οι προσπάθειες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ίσως να έχουν ως αποτέλεσμα μόνο ορισμένα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την υποστήριξη αυτή. Πρέπει να βρούμε λοιπόν το σωστό τρόπο αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί αυτή η πανευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού ίσως να είναι προς όφελος μόνο ορισμένων κρατών μελών. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, απλώς ε, να επισημάνω ε, ότι ήδη από τον τίτλο της πρότασης της Επιτροπής προκύπτει πόσο σημαντικό κομμάτι στην οικονομία της Ευρώπης παίζει ο τουρισμός επειδή αφορά και την πολιτική του. It's a new political framework for tourism. It's not just a framework, it's just a political framework. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η πρόταση δεν την έχω διαβάσει και ευχαριστώ πολύ την κυρία Ράνερ για την εισήγησή της, την πρώτη αυτή ενημέρωση, ότι είναι, έχει δύο σκέλη. Είναι η εξωστρέφεια, η Ευρώπη ως πόλος τουρισμού για τον κόσμο και η Ευρώπη και έχει μια ισοστρέφεια η Ευρώπη για τους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Από την άποψη αυτή αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται και το έχουν πει οι συνάδελφοι είναι μια καλή δικτύωση συνεργασίας και όχι ανταγωνιστικότητας με την κακή έννοια του όρου, συναγωνιστικότητας μάλλον και όχι ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στους τουριστικούς πόλους έλξης από τη μία μεριά και βεβαίως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αλλά πιστεύω ότι ήδη υπάρχουν οι θεσμοί όπως είναι οι πολιτιστικές διαδρομές όπως είναι το σήμα που ετοιμάζουμε να ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μπορούσαν από μόνο τους να αποτελέσουν αφορμή για μια τέτοια συναγωνιστική διάθεση. Εκτιμώ δηλαδή ότι είναι καιρός ως Επιτροπή Πολιτισμού, μιας και η, ε, η Κομισιόν και οι ε, Υπουργοί Πολιτισμού το, οι το έχουν καταλάβει στο ανώτατο επίπεδο, ότι είμαστε υποχρεωμένοι και ίσως έχουμε τρόπους να ζητήσουμε έξτρα χρηματοδότηση για την εφαρμογή τέτοιων δράσεων που στην ουσία υποστηρίζουν ακριβώς το πολιτικό πλαίσιο αυτή εδώ του, ε, αυτής εδώ της πρότασης. Εκτιμώ λοιπόν ότι του χρόνου θα πρέπει να απαιτήσουμε περισσότερα όχι μόνο για τις πολιτιστικές διαδρομές αλλά και για το σήμα και για άλλες δράσεις που πρέπει να ενταχθούν ωστόσο σε μια, ε, σε μια οργανωμένη ενότητα. Έχουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρουμε για το Eden χτες για παράδειγμα. Ξέρουμε όμως μερικά για τα, για τα cultural roots. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να οργανωθούν, να καταγραφούν όλες οι πολιτιστικές δράσεις που έχουν σχέση με τον τουρισμό και αυτό είναι νομίζω μια δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η Επιτροπή η δική μας και όχι κάποιος άλλος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Ράνερ και να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Μέρα Τουρισμού αφιερώθηκε στον τουρισμό εδώ χτες. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Εδώ δίπλα στην Επιτροπή και ο Επίτροπος για τον Τουρισμό και ο Επίτροπος για τον ε, Πολιτισμό είναι το ίδιο άτομο και αυτό είναι ένα δείγμα πολύ σημαντικό γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο ένα ταξίδι, μόνο το ταξίδι και η διαμονή. Ε, ξεπερνάει δηλαδή την Επιτροπή Μεταφορών. Ε, νομίζω ότι ε, εμείς, επαναλαμβάνω, είμαστε η πιο σημαντική Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Άρα θα πρέπει να τα να ξανασκεφτούμε τα θέματα. Θα πρέπει και εσείς, Πρόεδρε, κάτι να κάνετε για να επανέλθει μια ισορροπία, αν θέλετε, και να γίνει μια νέα κατανομή των αρμοδιοτήτων. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, στις τρεις βασικές στρατηγικές, στις τρεις βασικές στρατηγικές αναφέρει την ε, συλλογική προσέγγιση. Ο πολιτισμικός ο τουρισμός είναι ο πιο μεγάλος τομέας τουριστικός στην Ευρώπη και η Ευρώπη είναι ο πρώτος προορισμός στον κόσμο και λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα των, όλων των χωρών, ο πολιτισμός τελικά είναι το, ο καθοριστικός παράγοντας για να διατηρήσουμε αυτή την πρώτη θέση, την Γι' αυτό συμφωνώ κατά πολύ με αυτά που είπε η κυρία Ράνερ, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποια βασικά θέματα, για να επαναλάβουμε ακόμα και την, την κεντρική θέση που πρέπει να έχει ο πολιτισμός στον τουρισμό. Ε, Έχουμε υποβάλει μια τροπολογία στην Επιτροπή Προπολογισμού και ελπίζουμε θα περάσει για, μια, για ένα τριετές πρόγραμμα για, την, για τα τουριστικά, τις τουριστικές διαδρομές, γιατί εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε διακρατικά project, ούτως ή άλλως οι διαδρομές υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διακρατική συνεργασία, να, να αναπτυχθούν οι περιοχές αυτές και να προωθήσουμε ένα νέο τύπο τουρισμού τουρισμό. Διότι ο πολιτισμικός τουρισμός είναι το μόνο αγαθό το οποίο δεν μειώθηκε στον, αυτή την, περίοδο της κρίσης. Δύο πράγματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει στην γνωμοδότησή μας να υποστηρίξουμε την θέληση, τη θέλησή μας να υπάρχει αυτή η συλλογική η προσέγγιση ε, σε έναν διακρατικό τουρισμό Δεν ξέρω αν το, το τι θα είναι τέλος πάντων, τι θέλει να κάνει το Ευρωπαϊκό, αλλά τέλος πάντων ξέρω ότι στην Ιταλία μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι ε, ε το πόρταλ για, για τους Φραγκισκανούς που ξεκινάει από τον Κατέρμπουρη, φτάνει στην Ιταλία και μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Τέλος πάντων, ε, θα πρέπει να υλοποιήσουμε και να, να, μάλλον να εκπονήσουμε και να υλοποιήσουμε μία στρατηγική για τον τουρισμό. Ε, επίσης, ε, τα επαγγέλματα, τα τουριστικά επαγγέλματα πρέπει να τα προωθηθούν. Και πιστεύουμε ότι το πολιτισμικός ο τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός είναι στα χρόνια της κρίσης ένα μέσο για να ξεπεράσουμε την, τα προβλήματα θα πρέπει επίσης ο τουρισμός να ισχύει για όλες τις εποχές και για τις τέσσερις εποχές, όχι μόνο το καλοκαίρι. Χτες ε, ένα κορίτσα, ε, μια, μια κοπέλα, ε, Χριστίνα, ε, τρία-τρεις μήνες περπατούσε, ε, το μονοπάτι του, των Φραγκής ε, και βλέπουμε ότι, αυτό είναι μια ιστορία τώρα που σας λέω τέλος πάντων, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τέτοιου είδους προτεραιότητες για τους νέους. Επίσης το Next είναι ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν ε, ε, διάφοροι φορείς στην ε, Τοσκάνη για να συντονίσουν την τουριστική προσφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Ράνερ. όπω ε, και πολλοί προλαλήσαντε συνάδελφοι, έτσι και εγώ νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ανόητη ιδέα να αναλάβουμε εμεί ε, στην Επιτροπή μα τον τουρισμό. Στην Ισπανία, από τις αυτόνομες ε, περιφέρειες, 7 ή 8 έχουν αρμοδιότητα στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού. Υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν ε, παραλίες, δεν έχουν ε, θάλασσα. Εγώ πάντως ήμουν ε, περιφερειακός υπουργός για τη Μαδρίτη στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού. Δεν έχει θάλασσα, όπως ξέρετε, η Μαδρίτη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άλλα θέματα. Η Μαδρίτη προσελκύει μια εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, περισσότερους από χώρες άλλες. Άρα υπάρχουν αυτές οι αυτόνομες περιφέρειες που δεν έχουν θάλασσα ή άλλα αξιοθέατα τέτοια τουριστικά, αλλά έχουν ε, τους αντίστοιχες αρμοδιότητες. Και υπάρχουν πάρα πολλά ε, ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και μπορούν να ρυθμιστούν. Νομίζω ότι μπορούμε να ενώσουμε τους Ευρωπαίους, τους νέους με το Interrail. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, συνταξιούχοι που έχουν όλο και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Σίγουρα κυρία Πρόεδρε, όπως είπατε είναι δύσκολο να αλλάξουμε τις ημερομηνίε των διακοπών μας, αλλά με αυτές ε, τις ε, πτήσεις low cost μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και κάποια Σαββατοκύριακα για να πάμε ένα ταξίδι σε μια χώρα. Όπω είπε και η Σαμπίνε, δεν έχουμε μόνο την ε, κληρονομιά, αλλά έχουμε και κάποια θεάματα. Έχουμε τον τουρισμό που κάποιος πάει να επισκεφθεί διάφορα ωραία τοπία, για παράδειγμα. και επίσης ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ε, πολιτιστικό κυρίως τουρισμό ως ένα μέσο για να ενώσουμε τους Ευρωπαίους. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια στον τομέα αυτό και ίσως μια υπόδειξη προς ε, την Πρόεδρο είναι να προσπαθήσουμε να πάρουμε την αρμοδιότητα του τουρισμού στην Επιτροπή μας γιατί σχετίζεται άμεσα με πολλά από τα θέματα που μας απασχολούν εδώ. Tisztelt eh, kollégák! Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρατε για το Σιμπίου και τα χωριά εκεί πέρα γύρω, το Σιμπίου που ήταν ε, βεβαίως και πολιτιστική πρωτεύουσα και αύριο πάμε και στο ΠΕΤΣ, μια άλλη πολιτιστική πρωτεύουσα στην Ουγγαρία και εγώ θα τόνιζα και την, ε, το πώς μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά μέσω του πολιτισμού. Ξέρουμε πως υπήρχε το σιδηρούν παραπέτασμα που χώριζε την Ευρώπη σε ανατολική και δυτική, οπότε για μένα είναι απόλυτη προτεραιότητα η ανταλλαγή μεταξύ Ανατολής και Δύσης, να υπάρχει τουρισμός αμφίδρομος. Με φαντάζεστε πόσο σημαντικό είναι για κάποιον από την Ρουμανία να μπορεί να πάει στη Δύση. Επί δεκαετίες δεν μπορούσε να πάει στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή. Ε, γιατί πολλοί θεωρούν πως ε, η χώρα μας είναι μόνο Δράκουλας, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μνημεία εκεί πέρα. Και πράγματι έχουμε και ένα άλλο δρομολόγιο το οποίο θα μπορούσε να ανακαλυφθεί και αφορά και αιματικά λουτρά αλλά και μεταλλικά νερά. Το 1990 δε ιδρύθηκε και ένα πανεπιστήμιο εκεί στην ε, περιοχή το οποίο διδάσκει τα τουριστικά και θα θέλαμε βεβαίω να αναπτυχθεί και ο εκκλησιαστικός τουρισμός. Ε, είναι και αυτό σημαντικό να έρθουν πιο κοντά τα διάφορα δόγματα. Και ο διάλογος μεταξύ των δογμάτων είναι σημαντικός, αλλά και ο τουρισμός όπως σας είπα στα χωριά, στην Ήπεθρο Εάν γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον και αν θέλουμε να γνωρίσουμε ο ένας ε, τον άλλον πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως αυτό συνεισφέρει στο να πέσει και το συγκεκριμένο παραπέτασμα που υπάρχει στο μυαλό. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θεωρώ πως η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μας προσφέρει όχι μόνο την ευκαιρία αλλά και την υποχρέωση να ενισχύσουμε τον τουρισμό στην Ευρώπη γιατί έχουμε αυτό το οποίο θα έλεγε κανείς ε, αρμοδιότητες τώρα και οι οποίες είναι στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες. Ε, λοιπόν, πολιτικός τουρισμός, ο πνευματικός τουρισμός που θα συνδυάζεται με κάποιες δραστηριότητες όπως στο Σαντιάγο de Compostela και βεβαίω το να υπάρχουν ε, σύνδεσμοι μεταξύ των διαφόρων μέρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ αποφελές. Βεβαίω πρέπει να τονίσουμε πως το τουρισμός δεν είναι πολυτελή, είναι σχεδόν δικαίωμα. Και ειδικά με έναν πληθυσμό ο οποίος θα γυράσκει. Έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία να αναπτύξουμε στρατηγικές για να ενθαρρύνουμε όχι μόνο τους ανθρώπους να πάνε διακοπές, τους πιο ηλικιωμένους, αλλά να επεκτείνουμε και την τουριστική σεζόν, γιατί θα είναι ελεύθεροι να πάνε διακοπές ε, σε άλλες εποχές που οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές δεν θα μπορούν. Οπότε όσο περισσότερα κάνουμε εδώ πέρα, τόσο το καλύτερο. Και οτιδήποτε εξοδέψουμε στον τουρισμό βεβαίως θα αποδώσει σε δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου στις περιοχές εκείνες. Δεν συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή που είπε πως ε, κάθε χώρα πως επειδή κάθε χώρα δεν είναι εξίσου ελκυστική δεν αναπτύσσουμε πολιτική. Αυτή η λογική δεν εφαρμόζεται, δεν μπορεί να ισχύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχαμε αυτή τη λογική, παραδείγματο χάρη στου αυτοκινητόδρομου τη θαλάσση, δεδομένου ότι κάποιε χώρε έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στη θάλασσα από άλλε δεν θα έπρεπε να απτυχθεί τέτοια πολιτική. Πρέπει να δούμε λοιπόν το γενικό καλό. Και νομίζω πως κάθε χώρα έχει κάτι το ελκυστικό. Και κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάνε σε διαφορετικέ χώρε. Γιατί όλε είναι μοναδικέ. Και τέλος, να πω πως στη δική μου χώρα δυστυχώς είχαμε πτώση του τουρισμού από τη ΣΥΠΑ από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με μεγάλη αύξηση στον τουρισμό από την υπηρετική Ευρώπη. Και οι Ιρλανδοί που πάνε στο εξωτερικό τώρα κατευθύνονται και αυτοί στην υπηρετική Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν πως υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια θεώρηση της Ευρώπης ως μιας μονάδας και πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της ιδέας ότι θέλουμε μία Ευρώπη και ότι η Ευρώπη είναι ένα μέρος στο οποίο μπορούμε να προσελκύσουμε τουρίστες και απ' έξω βεβαίως από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά ιδιαίτερα από τον τουρισμό εντός της Ευρώπης. Και νομίζω πως έχουμε μια ευκαιρία, μια υποχρέωση θα έλεγα να διασφαλίσουμε πως πρέπει να το μεγιστοποιήσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Είναι καλό το ότι έτσι, προσπαθήσατε να πείτε και κάτι διαφορετικό στον κύριο Μεγκάλσκι. Κύριε Μεγκάλσκι, ε, ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν υφίσταται, αλλά υπάρχουν ε, πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί, πολλοί εντός της Πολωνίας, εντός της Γερμανίας και θέλουμε ακριβώς να αναδείξουμε αυτή την ποικιλομορφία. Θέλουμε να μάθουμε πώς είναι τα πράγματα στην Πολωνία, να μάθουμε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στη Βόρεια, στη Νότια Ρουμανία πώς είναι στο Κντάνσκ στην Κρακοβία, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Στο Βάτσλαφ που θέλουμε να πάμε. Οπότε παρεξηγειτε δεν θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε κάτι, να αναδείξουμε θέμε την ποικιλία, αυτή είναι η αποστολή μας. Και οι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έχουν βρει τον μπροστά του. Εμείς θέλουμε να τους αναδείξουμε όλους. Αυτό θέλουμε. Να ε, διατηρήσουν την αξία τους όλοι οι πολιτισμοί και να δούμε βεβαίω πράγματα που δεν είχαμε δει ως σήμερα. Μην είστε τόσο απεσιόδοξος. Δεν είμαστε οι κακοί εμείς εδώ πέρα. Θέλουμε αυτό το οποίο θέλετε κι εσείς να διαδώσουμε τον πολιτισμό. Οπότε Νομίζω πως εξαντλήσαμε το θέμα. Υποθέτω πως η κυρία Ράνερ άκουσε τα όσα είπαμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην... στο κείμενό σας. Περνάμε σημείο 12. Έχουμε μια μελέτη για το θέμα η συνθήκη τη Λισαβόνα και η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του αθλητισμού. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή και ελπίζουμε να μας πει και κάποια πράγματα η Κομισιόν και να ακούσει κάποια πράγματα για το πρόγραμμα του αθλητισμού το οποίο αναμένουμε για να εμπλουτιστεί και να βελτιωθεί. Οπότε έχουμε εδώ πέρα το ζητήσαμε αυτό, σε επιτροπή ζητήσαμε γνώμονες και στις 18 Νοεμβρίου έχουμε και μία ακρόαση στην οποία θα θέσουμε και ερωτήσεις θα προκύψουν από το κείμενο. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον κύριο καθηγητή Πάρης ο οποίος ήρθε μαζί με τον κύριο Μπόρχα Γκαρσία για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Έχουμε προβλέψει μία ώρα αλλά θέλω να σας παρακαλέσω να είστε ως δυνατόν πιο σύντομοι αλλά και ενδιαφέροντες. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Πάρης. Παρακαλώ κύριε καθηγητά. The pupils in the second row, please. Chair, thank you very much. Uh, thank... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Ο στόχος μας ε, είναι να κάνουμε μία μελέτη για τις ε, δυνατότητες ε, ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον αθλητισμό μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Καταρχάς σημειώσαμε ότι λέγεται ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της ε, ε, δίνει η συνθήκη. Και μέχρι να τεθεί ε, σε εφαρμογή η συνθήκη για τη λειτουργία της συνθήκης πέρυσι το Δεκέμβριο, δεν αναφερόταν αυτή η υποστήριξη. Αυτό δημιούργησε δύο βασικές ανησυχίες. Η πρώτη ήταν ότι η πολιτική για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό μέχρι σήμερα ε, καθορίζεται από, τα, από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και η νόμοι για την ενιαία ιστορική αγορά, δηλαδή η ελευθερία κινήσεων και αντα, ε, πολιτική ανταγωνισμού, δεν με την ιδιαίτερη σημασία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού. Η δεύτερη ανησυχία ήταν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική αθλητισμού ε, δεν έχει συνοχή και δεν έχει κύρος, διότι ακριβώς η ευρωπαϊκή ε, κοινότητα δεν είχε την άμεση αρμοδιότητα να χαράξει αθλητική πολιτική. Υπήρχαν κάποια ε, η, Κομισιό ε, έκανε κάποιες προτάσεις που αφορούσαν αθλητισμό, αλλά μέσα στα πλαίσια των ισχυουσών αρμοδιοτήτων, π.χ. για την πολιτική εκπαίδευση. Έπρεπε επομένως να δούμε κατά πόσον ε, οι νέες αρμοδιότητες που δίνει το άρθρο 165 συνθήκης ε, της Λισαβόνας παρέχει νέες αρμοδιότητες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν και θέματα ορισμού Δηλαδή, η, τι σημαίνει ευρωπαϊκή πολιτική αθλητισμού, τι, ποια είναι η ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, ε, τι σημαίνει να προωθήσουμε την ευγενή άμυλα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό κτλ. Όπως επίσης και τα θέματα της προστασίας της φυσικής και ηθικής ακαιρεότητας των αθλητών και αθλητριών στην Ευρώπη θα ασχοληθώ με το πρώτο θέμα, την πρώτη ανησυχία μας δηλαδή, ότι η εφαρμογή ε, των νόμων ε, που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και την ανταγωνιστικότητα δεν έλαβε υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού. Το άρθρο 165 θα οδηγήσει σε μια πιο συμπαθητική, αν θέλετε, εφαρμογή των κανόνων αυτών. Καταρχάς δεν υπάρχει ε, οριζόντια ρήτρα που να λέει ότι τα θέματα αθλητισμού και τα θέματα ευγενούς άμυλες ε, να λαμβάνονται υπόψη στην άσκηση άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπει η συνθήκη. Παραδείγματος χάρη ελεύθερη κυκλοφορία και ε, νόμος ανταγωνισμού. Και αυτό θα πρέπει να συγκριθεί με άλλες το, άλλους τομείς συνθήκης όπως ας πούμε η προστασία του περιβάλλοντος. Όπως όμως έδειξε και η απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση Μπερνάρ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Κομισιό, από ό,τι φαίνεται, δεν θα λάβουν υπόψη το άρθρο 165 υπόψη τους. Αυτό από καθαρής θεσμικής πλευράς δεν είναι σωστό. Εμείς πιστεύουμε ότι η η λήψη, το, το να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλητισμού είναι ζωτική σημασία για την εφαρμογή των, ε, ε της νομοθεσίας αυτής και αυτό πριν και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για τα αθλητικά, να, να δώσουμε στα αθλητικά σώματα ένα μεγάλο περιθώριο εκτίμησης είναι ουσιαστικό. Έστω και αν το άρθρο 165 δεν ε, επιβάλλει μία απέτηση να λαμβάνουμε υπόψη μας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλητισμού. Εμείς υποστηρίζουμε αυτό βλέποντας την ομολογία του δικαστηρίου και την, ε, τον τρόπο που λειτουργεί η Κομισιό από το Rave, από την υπόθεση ε, Wallrave μέχρι την υπόθεση Bernard πιο πρόσφατα. Όμως, ενώ είναι σωστό ότι η εξαίρεση, η αθλητική εξαίρεση που προβλέπεται στο Wall Rave στην υπόθεση Wall Rave έχει περιοριστεί σημαντικά από την πρόσφατη νομολογία, πιστεύουμε ότι και η ίδια αυτή η νομολογία δημιούργησε νέους δρόμους έτσι ώστε να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό του αθλητισμού και αναφέρομαι στους ε, στο δόγμα των εγγενών κανόνων που αναφέρονται στις υποθέσεις Μεντίνα. Επίσης, υπάρχει και ένα, ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Παραδείγματο χάρη στην, στα θέματα αντικειμενικών κριτηρίων και στα κριτήρια εξαίρεσης στον τομέα ανταγωνισμού. Θα δώσω το λόγο τώρα στον ε, συνάδελφό μου, τον κύριο Γκαρσία, ο οποίος θα ασχοληθεί με το δεύτερο θέμα το οποίο άφηξε στην εισαγωγή μου. το λόγο, παρακαλώ. Richard, thank you. Ευχαριστώ, Ρίτσαρτ. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω τώρα λοιπόν το δεύτερο μέρος της μελέτης μας, το οποίο αφορά το καθεστώς και την συνεκτικότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού ε, μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ο Δ. Πάρης σας ανέφερε τις βασικές ανησυχίες. Το κατά πόσον δηλαδή αυτό το νέο άρθρο μπορεί να ε, δώσει μεγαλύτερη συνέπεια και συνεκτικότητα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού. Αυτό αναλύσαμε λοιπόν στη μελέτη μας. Η ερευνητική ομάδα Κλήθηκε επίσης να εξετάσει πιθανούς τομείς δράσης ε, για την ε, πολιτική της Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού από το άρθρο 165 και θα κάνω και μία ε, σύντομη αναφορά και σε αυτό. Νομίζω ότι το πρώτο σημείο σε αυτό το δεύτερο τμήμα είναι ότι τώρα με την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα η πολιτική πια μπορεί άμεσα να εστιάσει στα θέματα του αθλητισμού χωρί να αναζητεί εναλλακτική νομική βάση όσο μεγαλύτερο ήταν ο αντίκτυπο, ε, μάλλον όσο μεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπο. όπως είπε ο κύριος θα είναι όχι στο νομικό, αλλά ε, στο αθλητικό κομμάτι. Δηλαδή θα έχουμε πιο συνεκτική πολιτική, αλλά βέβαια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τι προτάσει τη θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι το άρθρο αυτό απαιτεί να υπάρξει εστίαση στην ευρωπαϊκή διάσταση και ακριβώ να δικαιολογηθεί η προστιθέμενη αξία που θα αναλαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει δρομολογήσει με αυτή τη λευκή ε, βίβλο του 2007 μία συνεκτική πολιτική για τον τομέα του αθλητισμού, κάτι πολύ αναγκαίο και πρέπει αυτό να το εκτιμήσουμε. Το 165-4 ενισχύει τις προσπάθειες αυτές. Ε, κάτι πολύ σημαντικό που έχει σχέση με το νέο άρθρο είναι ότι τώρα η χρηματοδότηση των αθλητικών δράσεων είναι δυνατή χωρίς να πρέπει κανείς, όπως είπα, να αναφερθεί σε άλλες βάσεις ε, νομικές, που είναι δύσκολο να βρεθεί δυνατότητα χρηματοδότησης. Από όλους τους τομείς ε, πολιτικής θα αναφερθώ ακριβώς και σε αυτό το τομέα της εξέβρεσης χρηματοδότησης. Για να υπάρξει συνεκτικότητα στην πολιτική πρέπει να τεθούν σαφή στόχοι και σαφείς τομείς προτεραιότητας. Και αυτό πρέπει να γίνει ευθύς εξ αρχής. Γιατί αυτό θα διευκολύνει και την ε, εξέταση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής. Στη μελέτη μας λοιπόν συνιστούμε την ανάγκη καθορισμού μιας μικρής δέσου, πολύ σαφών προτεραιοτήτων για να υπάρχει αποτελεσματική δράση. Αναλύσαμε λοιπόν του τομεί προτεραιότητα στη μελέτη μας ε, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αφενό, λαμβάνοντα ε, το πλαίσιο τη διατύπωση του άρθρου. Μένουμε στη διατύπωση του άρθρου, τη συζητούμε, τη μελετούμε. Αφετέρου όμως είχαμε ε, και διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους φορείς, δηλαδή αθλητικές οργανώσεις, εθνικές κυβερνήσεις, κοινοβούλια, δηλαδή κυβερνητικού και μη κυβερνητικού οργανισμούς. Λάβαμε 37 περίπου απαντήσει από περίπου 50 διαφορετικές οργανώσεις. Κρατικέ και μη, όπω είπα. Τώρα, θα σας παρουσιάσω με αναλυτικό τρόπο τους τομείς πολιτικής, ε, μιλώντας και για το τι λέει το άρθρο και για τις προτεραιότητες των ενδιαφερομένων φορέων. Πρώτα απ' όλα, Υπάρχει ευρεία συμφωνία στο ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα για να έχουμε μια πολιτική βασισμένη στη γνώση. Έχει περάσει ο χρόνος ε, για να βασιζόμαστε σε υποθέσεις ε, στον τομέα του αθλητισμού, τα οποία δεν βασίζονται σε έρευνα και σε συγκεκριμένα πορίσματα. Και αυτό έχει να κάνει και με τα θεσμικά όργανα τη Ένωση και με τι αθλητικέ οργανώσεις που καλούνται τώρα να στηρίξουν τι αξιώσει του με έρευνα και με συγκεκριμένα δεδομένα. Οι οργανώσει αυτέ λοιπόν τώρα έχουν και αυτέ την ευθύνη να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη τη πολιτική αυτή. Του τομεί πολιτική και τι προτεραιότητε θα τι ε, υποδιαρέσω σε τρει ομάδε. Η πρώτη ομάδα είναι οι λεγόμενες ομόφωνες προτεραιότητες, γιατί πρώτα απ' όλα ευθυγραμμίζονται πάρα πολύ καλά με το άρθρο. Άρα εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα νομική βάση για την ανάπτυξη των πολιτικών αυτών. Δεύτερον, ευθυγραμμίζονται και με την τρέχουσα ημερήσια διάταξη, το τρέχον θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης και με τις ανάγκες και τις ε, απαιτήσει ε, των εμπλεκομένων φορέων. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, στόχος, πρόθεση καλών πρακτικών στον τομέα της ε, υγείας και της ε, σωματικής δραστηριότητας Φυσικά και θέλουμε να προωθήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωή σε όλη τη διάρκεια, σε όλο τον κύκλο ε, ζωή. Δηλαδή και για την νεολαία και για του ηλικιωμένους και αυτό σίγουρα σχετίζεται με τον τομέα τη εκπαίδευση, τη φυσική αγωγή και τη διδακτέα ύλη στα σχολεία. Δεύτερον, κοινωνική ένταξη και στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντάξουμε το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης στον αθλητισμό για να πετύχουμε μέσω του αθλητισμού την κοινωνική ένταξη. Και πρέπει να είναι σαφές αυτό. Δηλαδή συνιστούμε μια ολιστική προσέγγιση, η οποία, όπως ζητούν και κάποιοι ενδιαφερόμενοι φορεί, θα θίγει, θα αφορά κάποιες από τις πιο ε, μειονεκτικές ομάδες. Θέλουμε λοιπόν καταπολέμηση της ομοφυλοφοβία, καταπολέμηση της βίας, ισότητα των δύο φύλων. Τρίτη δέσμη στην ομόφωνη αυτή κατηγορία είναι η προώθηση του εθελοντισμού που ουσιαστικά ε, είναι η προώθηση των εθελοντών, ε, η προώθηση της, ε, του ερασιτεχνικού αθλητισμού και εδώ θέλουμε μια προσέγγιση η οποία θα ενθαρρύνει τον εθελοντισμό σε επίπεδο ατόμων μεμονωμένων αλλά και την άρση των ρυθμιστικών εμποδίων. Αυτό είναι η πρώτη κατηγορία λοιπόν ως τομείς προτεραιότητας. Δεύτερη ομάδα τώρα σχετική συμφωνία που δεν βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει πρόβλημα με την νομική βάση, ευθυγραμμίζεται καλά δηλαδή με το άρθρο και με το θεματολόγιο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, αλλά αυτές οι προτεραιότητε δεν ε, συμφωνούν με αυτές όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που μα απάντησαν. Στόχο εδώ λοιπόν είναι η διευκόλυνση τη έρευνα στον τομέα τη φαρμακοδιέγερση, του ντόπινγκ, αυτό είναι ένα ευαίσθητο, ένα λεπτό θέμα. Ε, έχει να κάνει με τις αθλητικές οργανώσεις. Υπάρχει, ε, υπάρχει ένα διεθνές πλαίσιο από τη Γουάντα, από την UNESCO και από το Ολυμπιακό κίνημα φυσικά. Αλλά υπάρχει ευρώ παιδί εφαρμογή, υπάρχει αίτημα για ευρωπαϊκή δράση, ιδίω για την εστίαση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, σε ό,τι αφορά το ντόπινγκ, βελτίωση επίδοση, σχετικά φάρμακα, σε γυμναστήρια κτλ. Και ίσω υπάρχει και το αίτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει το συντονισμό της έρευνας και το συντονισμό μεταξύ των εθνικών οργανισμών καταπολέμησης του ντόπινγκ. Δεύτερο, σε αυτή τη δεύτερη ομάδα, ενθάρρυνση ενός κοινωνικού και δομημένου διαλόγου στον τομέα του αθλητισμού. Εδώ το πρόβλημα ίσως είναι ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Εμείς πάντως θεωρούμε ότι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου είναι κλειδί για την καλή διακυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν ενθαρρύνουμε τον κοινωνικό διάλογο υπό την αιγίδα βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τρίτη δέσμη προτεραιοτήτων, τρίτη ομάδα ετοιμάτων ίσως αν θέλετε, που όμως θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να συσταθούν γιατί δεν συμφωνούν με το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως είναι δύσκολο να λάβουν θετική νομική γνωμοδότηση. Έγκριση λοιπόν κατευθυντηρίων γραμμών, την εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στον τομέα του αθλητισμού. Νομίζουμε ότι οι κατευθυντήριε αυτέ γραμμέ δεν θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στον τομέα του αθλητισμού. Και δεύτερο, σε αυτή την τρίτη και τελευταία κατηγορία, ε, ω αίτημα είναι ο ορισμό τη ε, ιδιαιτερότητα, του specificity. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ορισμό τη έννοια αυτή και όπω είπε και ο Δόκτωρ Πάρη, οι αθλητικοί φορεί τώρα πρέπει να αναλάβουν προβλεπτική δράση. Υπάρχει η αρχή τη καλή διακυβέρνηση και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να ε, καθορίσουν από μόνοι τους αυτή την specificity, αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτά σε ό,τι αφορά ε, το καθεστώς και τώρα συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εννέα πολύ συγκεκριμένα σημεία για να συνοψίσουμε τα 50, τις 50 σελίδες της μελέτης μας. Πρώτον, το άρθρο 165 δεν περιέχει μια οριζόντια ρήτρα. Επομένως, η αναφορά στην ειδική φύση, στον ειδικό χαρακτήρα του αθλητισμού, νομίζουμε ότι μάλλον θα επηρεάσει το δικαστήριο και την Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχει συνταγματική ανάγκη και συνταγματική υποχρέωση να ληφθούν υπόψη διατάξει αυτέ. Δεύτερο, νομίζουμε ότι η εκπώνηση κατευθυντηρίων γραμμών ε, για να μεταφερθούν κανόνε ανταγωνισμού στον αθλητισμό ίσω να μην βοηθήσει τόσο πολύ την ε, επιδίωξη ε, της ασφάλειας δικαίου, γιατί ο ειδικό, ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού αναγνωρίζεται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, οι αρμόδιοι αθλητικοί φορείς θα πρέπει να αναλάβουν τον ορισμό της ιδιαιτερότητας στο πλαίσιο της αρχής καλής διακυβέρνησης. Τέταρτον, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την εθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα ε, του αθλητισμού και θα πρέπει ε, και ο δομημένος διάλογος να μην, ε, να μην υπονομεύσει αυτή την προσπάθεια. Πέμπτον, ο δομημένος διάλογος είναι ή μπορεί να είναι προβληματικός λόγω της ποικιλομορφία του αθλητικού κινήματος. Γι' αυτό λοιπόν συνιστούμε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην πιστεύουν ότι μία μεμονωμένη δράση μπορεί να εκπροσωπεί τον κόσμο του αθλητισμού εν γέννη, γιατί είναι μεγάλη ποικιλία και ποικιλομορφία. 6. Το άρθρο 165 επιλύει ζητήματα νομικής ε, ασάφειας για κάποια προγράμματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό. 7. Θα πρέπει να προτιμηθεί μια μικρή δέσμη προτεραιοτήτων. 8. Θα πρέπει η χάραξη πολιτικής να βασίζεται σε συγκεκριμένες αποδείξεις, να είναι evidence-based και θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να δικαιολογούν τις θέσεις τους με στέρεα στοιχεία και έρευνα. Και τέλος, ένα το σημείο, υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς πολιτικής που συγκεντρώνουν μεγάλο βαθμό ομοφωνίας. Εκπαίδευση, υγεία και σωματική άσκηση, κοινωνική ένταξη στον αθλητισμό, ώστε να πετύχουμε την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού και τρίτο, προώθηση του εθελοντισμού. Αυτές λοιπόν είναι και οι βασικές ε, γραμμές, τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε και μια σύνοψη της έκθεσης στον φάκελό μας. Εάν δείτε στα εγγραφά σας υπάρχει μια σύνοψη της μελέτης. Αν δεν θέλετε να διαβάσετε ολόκληρη, πάρτε τουλάχιστον τη σύνοψη, είναι πολύ σημαντική. Και την έχουμε και τυπωμένη την ίδια τη μελέτη και θα εμφανιστεί και στην ιστοσελίδα στα αγγλικά πρώτα και μετά στις υπόλοιπες γλώσσες. Στο site που αναφέρεται εδώ πέρα. Τώρα λοιπόν, κυρία Καμαγεβέτη, να ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Ε, είναι ενθαρρυντικά αυτά τα οποία που ακούμε, αλλά από την άλλη και κάπως απογοητευτικά γιατί έχω την εντύπωση πως ε, νομίζω πως ε, μας είχαν υποσχεθεί περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε με το άρθρο 165. Να πω ένα παράδειγμα μόνο, εάν κατάλαβα καλά. Προειδοποιήσατε για το αν θα πρέπει να δημιουργούμε πανευρωπαϊκές νομικές βάσεις. Και εδώ πέρα εμείς είχαμε υιοθετήσει μεγάλη πλειοψηφία, ένα ψήφισμα για τους ε, μάνατζερ ε, παιχτών. Και αυτό ακριβώς ανταποκρίνεται σε αυτό το νομικό πλαίσιο και εγώ είχα συναντηθεί ε, με έναν εκπρόσωπο, τον μάνατζερ, τον μάνατζερ σωστά, των παικτών του χόκεϊ, αλλά αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα αθλήματα. Και μου είπε, μακάρι να είχαμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα διοδότησης των μάνατζερ των παιχτών. Ε, τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο σύστημα, γιατί κάποιο είναι στη Γερμανία, πρέπει να πάει σε άλλο σύνδεσμο να εγγραφεί στην Αυστρία και είναι πολύ πλοκο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα το οποίο θα είναι νομικά δεσμευτικό και το οποίο βεβαίως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι ανοιχτό σε προσφυγές και δεν είναι δίκαιο αυτό και για τις ομάδες και για τους παίκτες αυτή η ασάφεια δικαίου. Και εμείς ως Κοινοβούλιο λέμε θα θέλαμε να κάνει κάτι η Κομισιόν, να έχουμε μια νομική βάση και ένα τέτοιο σύστημα διοδότησης. Λέτε καλύτερα λοιπόν να μην κάνουμε τίποτα γιατί δεν υπάρχει η νομική βάση. Οπότε υπάρχει κάποιος διχασμός, αν θέλετε, όσον αφορά το αποτέλεσμα της ε, μελέτης σας. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα μια σύγκρουση, αν θέλετε, του δικαίου του ανταγωνισμού και του δικαίου της εσωτερικής αγοράς. Και να δούμε τι θα κάνουμε μέσω του άρθρου 165 για να δημιουργήσουμε περισσότερη συνεκτικότητα και ασφάλεια του δικαίου, ειδικά τουλάχιστον για τους επαγγελματίες αθλητές. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Ναι. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή Πιστεύω ότι ο αθλητισμός, όπως είπατε και εσείς πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας και σας συγχαίρω κυρία Πρόεδρε για τον ενθουσιασμό σας ε, για αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει καταρχάς να στοχεύουμε σύντομες νίκες και σε τρεις τομείς μπορούμε να έχουμε αυτές τις σύντομες νίκες και, μεγάλες, ε, και μεγάλη συνεισφορά. Κοινωνική συνοχή, ε, εθελοντισμός και ε, αθλητικές δραστηριότητες, γυμναστική. Και πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθούν όλες αυτές οι δράσεις στην Ευρώπη. Σε σχέση με τον εθελοντισμό, θα ήθελα να ρωτήσω μία ερώτηση. Είπατε ότι Υπάρχουν ε, κάποια κανονιστικά εμπόδια στον εθελοντισμό. Ποια είναι αυτά και πώς μπορούμε να, το, να τα καταργήσουμε. Για τον ντόπινγκ επίσης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή το, το, το ντόπινγκ δεν έχει τόση μεγάλη σημασία όσο είχε πριν από μερικά χρόνια. Και ίσως να υπερβάλλουμε. Δηλαδή, ένας υπέας, ο ένας τζόκι πριν από μερικές εβδομάδε, ο οποίος πριν από τη συμμετοχή του σε κάποιες υποδρομίες, μία Παρασκευή πρωί, έκανε, πέρασε από τέστε και του είπαν ότι έχει διπλά, διπλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και δεν έπρεπε να πάρει μέρος αγώνες. Αυτός όμως δεν είχε πιει ούτε μία σταγόνα για 15 χρόνια. Και Α, και τελικά το αποτέλεσμα ήταν, ε, καταλάβανε, καταλήξαν στο συμπέρασμα, ότι βγήκε το τεστ, ε, είχε το τεστ αυτά τα αποτελέσματα, διότι είχε χρησιμοποιήσει ένα δοντικό διάλειμμα ο άνθρωπος για να πλύνει τα δάλια του το πρωί. Τέλος πάντων, πρέπει να δούμε πια, κάποια κανονιστικά μέτρα, τα οποία θα προστατεύσουν τους αθώους και θα βρίσκουν ταυτόχρονα και τους ενόχους. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, περιμένουν από εμά να κάνουμε πολλά πράγματα και είδαμε χτες ότι όταν συζητάγαμε ε, τα θέματα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσα του Αθλητισμού, ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε ένα χρονικό διάστημα και γι' αυτό πιστεύω ότι σε αυτές τις σύντομες νίκες πρέπει να ποντάρουμε πρώτα. Ευχαριστώ παρακαλώ να είστε λίγο σύντομοι, κύριε Μπόρις. Dziękuję bardzo za, za tę analizę. Ναι, όντω. για τον αθλητισμό δεν έχουμε δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό να νομοθετήσουμε. Αλλά το άρθρο 165 μας δίνει την δυνατότητα να παρέμβουμε στον, αθλητικό τομέα και πρέπει αυτός να είναι ο επόμενος τομέας στον οποίο θα νομοθετήσουμε στην Ευρώπη. Τώρα, καταρχάς έχουμε τα θέματα προ... προπόνησης, αν θέλετε, στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ε, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ καλά στην Ευρώπη. Βλέπουμε τους αθλητές που έρχονται από άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης, που και αυτό αποδεικνύει ε, ότι γενικά τα προπονητικά θέματα δεν πάνε καλά στην Ευρώπη. Ίσως, ε, επομένως, ε, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ίσως θα έπρεπε να δούμε και πόσο θα, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση για, τα, ε, για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Διότι, ας πούμε, οι διάφοροι αθλητικοί όμιλοι έχουν χρήματα, πολλά χρήματα στη διάθεσή τους, πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία χρειάζονται. Και δεν μιλάω μόνο για τους ποδοσφαιρικούς ομίλους. Ίσως θα έπρεπε κάπως να νομοθετήσουμε στον τομέα αυτό. Ivo Ehm, eh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις στα Ολλανδικά. Βεβαίως δεν είχα την ε, ευκαιρία να διαβάσω ακόμα τη μελέτη. Αλλά έχω την αίσθηση πως ε, είναι σαφής η δυνατότητα να κάνουμε κάποια πράγματα με το νέο αυτό άρθρο στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, της διαφοράς ε, στον αθλητισμό και μία ερώτηση προς τους ε, καθηγητές. Αν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την απάτη στο τύχημα, παραδείγματο χάρη, χρειαζόμαστε μία επιπλέον νομική βάση. Και δεύτερον, λέτε στα συμπεράσματα, με κάπως περίεργη διατύπωση, γι' αυτό θέλω μία διευκρίνηση, ε, υπάρχει ένα αίτημα για κατευθυντήριες γραμμές στον αθλητισμό και αν κατάλαβα καλά, λέτε πως αυτό δεν είναι καλή ιδέα να έχουμε κατευθυντήρες γραμμές γιατί είναι πολύ γενικές και θα αφορούν όλα τα αθλήματα μαζί, ενώ θα πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση. Και το ερώτημά μας ήταν, και αυτό το οποίο θέλαμε, είναι πάντα να φύγουμε από τη κατά περίπτωση αντιμετώπιση και να πάμε σε μια γενική αντιμετώπιση με μια έτσι νομική βεβαιότητα. Θεωρείτε πως αυτό δεν είναι επιθυμητό ή δεν είναι εφικτό έχετε κάποιε άλλε σκέψεις να μα προτείνετε. Ευχαριστώ, Σαντιάγκο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το άρθρο 165 αυτό που επιτρέπει κυρίως είναι η πολιτική βούληση για να ασχοληθούμε με το θέμα του αθλητισμού. Ίσως πριν να μην υπήρχε αυτή η νομική βάση. Γνωρίζω ότι είναι ένα περιοριστικό βέβαια άρθρο σε μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα όμως να ακούσω και την Κομισιόν η οποία θα πρέπει να δημοσιεύσει μια σχετική ανακοίνωση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αθλητισμό μέσω του άρθρου 165, αλλά και μέσω άλλων ενιών για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να δουλέψουμε. Ελεύθερη κυκλοφορία, ντόπινγκ, βία, στοιχήματα που ανέφερε η Βομπέλετ που έχουν να κάνουν το εσωτερικό, με την ιστορική αγορά, αρμοδιότητα του Επιτρόπου, Μπαρνιέ, διακριτική μεταχείριση, εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπορεί να μην ε, είναι άμεσα ε, εντασσόμενα στο άρθρο 165. Αλλά αν δούμε τι αρμοδιότητε του 165 συν τι άλλε αρμοδιότητε που μπορούμε να έχουμε από ε, άλλε πιο γενικέ αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ήδη ισχύουν, και κυρίως βέβαια αν υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί αυτό που είναι σαφές είναι ότι είναι μεγάλες οι προσδοκίες στον κόσμο του αθλητισμού. Και πρέπει να δουλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να επεξεργαστεί το θέμα αυτό. Και έτσι νομίζω ότι με όλα αυτά μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι πιο στέρεο, υπερβαίνοντα τι περιορισμένε αρμοδιότητε του άρθρου 165. Ευχαριστώ όσα ακούστηκαν, σύντομα μόνο. Θεωρώ πως πρέπει να ερμηνεύσουμε το άρθρο 165 για να έρθουν οι περισσότερες αρμοδιότητες του αθλητισμού στην Ευρώπη και θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, συντάκτες της έκθεσης αν είναι τα πράγματα πράγματι όπως ε, τα φοβούνται και να συμφωνήσω με την συνάδελφο εδώ πέρα. Πράγματι θα πρέπει να δούμε με τους ε, μάνατζερ εκεί πέρα να γίνει ένα πανευρωπαϊκό επάγγελμα και εντάξει για να μην μιλήσω τώρα για τις ελλείψεις του προπολογισμού εάν δεν έχουμε καν την ε, νομική βάση την ε, δυνατότητα να δραστηριοποιηθούμε το ερώτημα είναι το άρθρο 165 είναι τόσο μικρό και ανεπαρκές όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, σας ευχαριστώ. To our Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στους ε, προσκεκλημένους μας. Θεωρείτε πως η ΒΑΔΑ, η Παγκόσμια Ένωση, η καταπολέμηση του ντόπινγκ είναι το κατάλληλο πλαίσιο καταπολέμησης του ντόπινγκ. Ή χρειαζόμαστε μια εναλλακτική λύση. Η Ευρωπαϊκή λυση μια ευρωπαικη ενωση πολέμησης του ντόπινγκ. Ή κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Να συμφωνήσω και εγώ με τις απογοητευμένες κυρίες και εγώ απογοητεύτηκα. Έχω λοιπόν δύο συγκεκριμένα ερωτήματα για το θέμα των μάνατζερ των παικτών και την αδειοδότησή τους. Μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όχι. Αν όχι, δεν μπορούμε και, και να βοηθήσουμε εδώ πέρα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αυτό το οποίο έχουμε θέσει ως στόχο, δηλαδή να βρούμε μια ισορροπία στον μέτρο δεν θα τα καταφέρουμε. Δεύτερον, για το θέμα του οικονομικού fair play μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε Ήρθαν εδώ πέρα η UEFA, η FIFA και λένε θέλουμε βοήθεια. Θέλουν να τους βοηθήσουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε εμείς να την προσφέρουμε. Πρέπει να ερμηνεύσουμε τόσο στενά το άρθρο 165 ώστε να μπορούμε μόνο να μιλάμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα νομοθετικά, να βοηθήσουμε. δηλαδή και το θέμα ακριβώς χρηματοδότησης που αναφέρθηκε. Δίνουμε ένα των ε, χρημάτων που έχουμε. Αν δούμε π.χ. Τη, στήριξη του καπνού είναι επίσης 1%. Δηλαδή αναρωτιέμαι σε τι κοινότητα ζούμε. Δηλαδή από τη μία απαγορεύουμε παντού το κάπνισμα και εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν καπνίζω κιόλα. Οπότε το αντιλαμβάνομαι γιατί με ενοχλεί. Από την άλλη προωθούμε την καλλιέργεια του καπνού με 1% του προπολογισμού μας. Και για όλους τους τομείς μας ε, έχουμε επίσης 1%. Ε, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα θυμώσουν οι Έλληνες ε, ή ποιος άλλο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το, το θέμα, να το συζητήσουμε με τις κυβερνήσεις μας. Ε, δεν είναι ισορροπία αυτή. Λοιπόν, α, η Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Ποιος μπορεί να μας διαφωτίσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ήθελα καταρχάς ε, να χαιρετήσω τη μελέτη αυτή που ανάθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία θα δώσει τροφή στη φάση προβληματισμού και σύνταξης ε, των μελλοντικών πρωτοβουλίων της Κομισιόν στον τομέα αυτό από τη στιγμή που ο αθλητισμός αποτελεί μια νέα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι νέα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 165. Ωστόσο οι άλλε διατάξεις που μπορούν να επηρεάσουν τον αθλητισμό και υπάρχουν ε, ήδη στη συνθήκη εξακολουθούν να ισχύουν. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010, όπως τουλάχιστον έχουμε προγραμματίσει, θα δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για τη συνθήκη της Λισαβόνας και τον αθλητισμό. Σε αυτή την ανακοίνωση στόχος μας θα είναι να καθορίσουμε από τη δική μας ε, σκοπιά το πλαίσιο που πρέπει να διέπει τις μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα του αθλητισμού, οι οποίες θα υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρατηρώ ότι πολλά από τα στοιχεία τα οποία μας απασχολούν ε, βλέπω με χαρά ότι αναφέρονται στην έκθεση των ε, καθηγητών. Έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις που θα βοηθήσουν ε, την άσκηση προβληματισμού για την πρόταση αυτή και έχουμε διαβουλεύσεις ε, με τα κράτη-μέλη, τον Ευρωπαϊκό Φόρουμ που είχαμε στη Μαδρίτη, με τις ε, αθλητικές οργανώσεις, είχαμε μια ηλεκτρονική διαβούλευση, κάτι ριζοσπαστικό και δείχνει, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, δείχνει αυτό πόσο ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 1.300 συμβολείς, 1391 συγκεκριμένα αθλητικές οργανώσεις συμμετείχαν. Εξέφρασαν πολλές ε, διαφορετικές απόψεις, ε, πολλές ήταν υπέρ της αρχής της αυτονομίας και της επικουρικότητας. Επίσης, λάβαμε έγγραφα από διάφορες ε, αθλητικές οργανώσεις οι οποίες ανέφεραν συγκεκριμένα τις τοποθετήσεις τους. Επίσης, η κυρία Βασίλειο Αρμόδια Επίτροπος για να τροφοδοτηθεί αυτή η διαδικασία θέλησε να συγκροτηθεί μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με προσωπικότητες, άλλοι από την πολιτική, άλλοι από ε, τον κόσμο των πανεπιστημίων. Και ο κύριος Πάρης ε, που είναι ο επικεφαλής ε, της μελέτης, ο κύριος Μαυρομάτης, εξευωνίμων μου. Είχαμε λοιπόν αυτούς τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν μια ανεξάρτητη τοποθέτηση που θα τροφοδοτήσει της, ε, το, τη διαδικασία αυτή και την ε, επεξεργασία του θέματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, υπάρχει μια ακαδημαϊκή επιστημονική προοπτική. Τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να προταθεί με βάση το άρθρο αυτό το προβλεπόμενο στη συνθήκη, αλλά και με βάση άλλες διατάξεις της συνθήκης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς ε, τη μελέτη αυτή, τις προτάσεις τα συμπεράσματα και συγκεκριμένα την τελευταία παράγραφο της παραγράφου του σημείου 6. Θα ήθελα να πω στην Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτισμού ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη μελετά, ε, εξετάζει αυτή τη μελέτη, θα τη λάβει υπόψη, την είχαμε λάβει την προηγούμενη εβδομάδα, τη μελέτη αυτή, και σε μεγάλο βαθμό οι προτεραιότητες που εντοπίζει η μελέτη ως ε, προτεραιότητες σχετικές με την πρόθεση της φυσικής δραστηριότητας, σωματικής άσκησης δηλαδή, την κοινωνική ένταξη μέσω του θελοντισμού, είναι προτεραιότητες που και εμείς έχουμε συμπεριλάβει στην έγγραφα εργασία μας. Και ελπίζω όταν σας παρουσιάσουμε στα τέλη του έτους την ανακοίνωση για την οποία έκανα λόγο, να μπορέσετε κι εσείς να διαπιστώσετε ότι πολλά από τα στοιχεία τα οποία εντοπίζονται στη μελέτη τα έχουμε ήδη λάβει υπόψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ war nicht minder desillusioniert. Και αυτό ήταν κάπως απογοητευτικό. Κύριε Δελγάδο. Κύριε καθηγητά, κύριε Πάρης, είστε και εσείς σε αυτή την ομάδα των ειδικών. Εάν μας πείτε και εσείς τα ίδια, τα βλέπω μαύρα τα πράγματα. Αλλά απαντήστε στα ερωτήματα που ο Γκαρσία, παρακαλώ. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία εμπεριέχονται σε αυτές τις ερωτήσεις. Αυτό το οποίο θα πρότεινα είναι το εξής. Το πρώτο θέμα το οποίο αναδεικνύεται είναι τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τις δυνατότητες εναρμόνισης. Και ένα άλλος συνάδελφος θα ασχοληθεί με αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, ο κύριος Γκαρσία θα ασχοληθεί και τη τρίτη κατηγορία, αν θέλετε, θεμάτων, αν κατάλαβα καλά, έχει να κάνει με κάποια νομικά θέματα σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές, και την προσέγγιση ανά περίπτωση. Γι' αυτά θα μιλήσω εγώ. Ο κύριος Μίρτεν έχει το λόγο πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τα θέματα τα οποία έθεσε η Επιτροπή σας για τα θέματα αναρμόνισης και το άρθρο 165, Ήθελα να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι για το κατά πόσο μπορεί κανείς να νομοθετήσει σε αυτούς τους τομείς, αλλά για το κατά πόσο το 165 επιτρέπει να το κάνουμε. Το άρθρο 165 αναφέρει την ε, εναρμονισμένη πολιτική και το πρόβλημα είναι απαγορεύει το άρθρο 65 εναρμόνιση μεν, αλλά αυτή η εναρμόνιση απαγορεύεται και σε άλλους τομείς. Όχι, δεν το λέει αυτό το άρθρο, το άρθρο 165. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε άλλα, άλλη νομική βάση. Υπάρχει το άρθρο 114, α πούμε, για την, για την ενιαία εσωτερική αγορά. Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν νομική βάση. Τώρα, σαν αφορά το οικονομικό έγκλημα που θύχθηκε αυτό, εδώ το, η συνθήκη της Λισαβόνας ε, παρέχει ένα πλεονέκτημα, διότι μας επιτρέπει να νομοθετήσουμε σε τομείς όπου υπάρχουν διακρατικά στοιχεία, υπερεθνικά στοιχεία, αν θέλετε, εγκληματικότητας. Επομένως, στο θέμα της ε, εναρμόνισης και νομοθεσίας γενικά, η νομοθεσία για την ενιαία εσωτερική αγορά ε, ρυθμίζει πολλά πολλούς τομείς ε, του αθλητισμού και αυτούς που δεν ρυθμίζει μέχρι τώρα μπορούμε να τους ρυθμίσουμε στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ποια είναι η πλέον κατάλληλη νομική βάση. Όσον αφορά τώρα το κατά πόσον το 165 απαγορεύει την αναρμόνιση επειδή λέει ότι από μόνο του δεν επιτρέπει το άρθρο αυτό την αναρμόνιση ε, αυτό γίνεται με βάση την ομολογία για την δημόσια υγεία και για το τσιγάρο η νομοθεσία που απαγορεύει το κάπνισμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα μεν, αλλά ο φορέας για να γίνει κάτι τέτοιο, με μια πρώτη ματιά δεν φαίνεται να είναι το άρθρο 165. thank you. Ευχαριστώ, πολύ. Επειδή έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στη μητρική γλώσσα αυτό το καταπληκτικό εργαλείο της Διερμηνίας, θα το πράξω και εγώ, θα μιλήσω ισπανικά. Φυσικά και διακρίνω αυτό το αίσθημα απογοήτευσης ε, των βουλευτών της Επιτροπής σας για το τι μπορεί να γίνει και το τι δεν μπορεί να γίνει ή τι μπορούμε να νομοθετήσουμε και τι δεν μπορούμε. Πράγματι, νομοθέτες, τα κράτη-μέλη, στην κυβερνητική διάσκεψη όταν ε, εισήγαγαν αυτό το άρθρο το έκαναν σε επίπεδο πιο χαμηλό στο, στο κατώτερο μάλλον επίπεδο αρμοδιότητων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό είναι περιοριστικό και περιορισμένο στο πεδίο εφαρμογή του και το άρθρο αυτό. Ο Σάμιλ σας τα είπε και πριν πάντως εμείς παρόλα αυτά θεωρούμε ότι ανοίγει πόρτες αυτό το άρθρο. Και ίσως αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να αναφερθούμε και να εστιάσουμε στις πόρτες, στα παραθυράκια αυτά. Στα συμπεράσματά μας αναφέρουμε ορισμένους τομείς ε, στα συμπεράσματα μόνο, γιατί στην έκθεση ε, είναι πολύ περισσότεροι τομεί που αναφέρουμε. Στους τομείς πάντως που αναφέρουμε στα συμπεράσματα, στους πέντε αυτούς, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια προστιθέμενη αξία και να αναπτύξουμε μια πτυχή του, του αθλητισμού. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η πτυχή είναι αυτή η οποία ε, ενδιαφέρει περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο επαγγελματικό αθλητισμός ίσως προσελκύει ε, τους ε, αθλητές, έχουμε το οικονομικό fair play, αλλά όπως δείχνει το ευρωβαρόμετρο, ειδικά για τον αθλητισμό, οι Ευρωπαίοι ασκούνται, κάνουν αθλητισμό με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μιλάμε δηλαδή για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που γίνεται ενίοτε σε κάποια αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια κτλ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πτυχές κοινωνικές που σχετίζονται με τους πολίτες φαίνεται να υπάρχει μάλιστα συνένεση και μεταξύ όλων των ε, οργανώσεων του κλάδου ότι αναμφίβολα μια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να προσθέσει αξία, μεγάλη αξία και αυτό αφορά εκατομμύρια πολίτες. Δεν είναι λοιπόν κάτι αμεληταίο, δεν είναι κάτι ασήμαντο και τετριμένο. Τώρα, έρχομαι στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Για τα, τους φραγμούς κάποιος ρώτησε, για τα εμπόδια στον εθελοντισμό. Από ό,τι φαίνεται, από τη μια πλευρά φυσικά και ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο εθελοντισμός και υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά κυρίως εμπόδια. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι με το άρθρο 165 είναι δύσκολο να νομοθετήσει κανείς για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου. Απ' την άλλη όμως θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλες νομικές βάσεις στις οποίες θα μπορούσαμε να αναφερθούμε. Κάτι άλλο που μπορεί να βοηθήσει κανείς είναι αν μπορούμε να άρουμε τα εμπόδια τα οποία δημιουργούν οι ίδιες αθλητικές ομοσπονδίες για την ε, πρόσληψη, ε, για το, την ανάθεση καθηκόντων σε εθελοντές ε, κτλ. Ή διανομή, ε, διάδοση μάλλον, ε, η κοινοποίηση καλών πρακτικών για το τι μπορεί να γίνει, είναι καλό και αυτό. Και νομίζω ότι και η δική σας επιτροπή μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε έναν ε, τομέα που έχει τονιστεί σε μια έκθεση για τον εθελοντισμό. Δηλαδή υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ του τι θέλουν οι εθελοντές και το τι θέλουν οι οργανώσεις. Ο Ευρωπαϊκό Εθελοντισμό ιδίως στον τομέα του αθλητισμού, έχει να κάνει κυρίω με τη νεολαία. Είναι νέοι οι οποίοι ψάχνουν μια μικρή περίοδο εθελοντική εργασία. Οι οργανώσει όμω συνεχώ απαιτούν πιο πολλά πράγματα από του εθελοντέ του. Να είναι για πιο πολύ χρόνο, να έχουν πιο πολλέ ειδικέ γνώσει και δεξιότητε, δηλαδή και του αναθέτουν πολλέ ευθύνε και έχουν μεγάλε απαιτήσει από αυτού. Πρέπει λοιπόν να δούμε με τι οργανώσει αν θα μπορούσαν να αναπτύξουν τον εθελοντισμό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ανάγκες και οι προσδοκίες να μπορούν κατά κάποιο τρόπο να συμφιλωθούν μεταξύ τους και να συμπέσουν ώστε να ασχοληθούν όλο και περισσότεροι νέοι με τον εθελοντισμό. Μια άλλη ερώτηση που ετέθη ήταν η χρηματοδότηση των μάνατζερ, των ε, παικτών, των αθλητών εν γέννη. Αυτό το είδαμε στη μελέτη μας, ο Ρίτσαρτ Πάρις μπορεί να σας πει περισσότερα όταν λάβει το λόγο. Είναι κάτι το οποίο το μελετάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμιση. Εμεί στη μελέτη μας βλέπουμε ότι αυτό το οποίο μέχρι τώρα ήταν ένα αρκετά μεγάλο αίτημα από τον αθλητικό κόσμο, τώρα, τουλάχιστον στην περίπτωση ορισμένων μάνατζερ, δεν υπάρχει πια, έχει αποσυρθεί αυτό το αίτημα. Ίσως όμως καλό θα ήταν να υπάρξει ε, νομοθεσία σχετική. Τώρα, τι μπορεί να γίνει για τα στοιχήματα να μην υπάρχει τόση διαφθορά στο στοιχηματισμό. Υπάρχουν αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμοδιότητες συντονισμού στον τομέα στο χώρο μάλλον της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Υπάρχει συντονισμός των προσπαθειών ε, των ε, δυνάμεων ασφαλείας. Ε, και σε ό,τι αφορά τα γραφεία στοιχηματισμού σίγουρα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συνεργασία και μεταξύ κρατών μελών δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εναρμόνιση, δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή νομοθεσία, δεν μπορεί να νομοθετήσει κανείς και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Θα αφήσω όμως τον Ρίτσαρτ Πάρις να μιλήσει για την καταπερίπτωση αντιμετώπιση, για τις κατευθυντήριες γραμμές και τέλος να πω, απαντώντας ε, στο ερώτημα που αφορούσε την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πω το εξή. Κάθε φορέ όλο και περισσότερε φωνέ ακούγονται από τον ίδιο τον κόσμο του αθλητισμού και από τα κράτη-μέλη για την αναποτελεσματικότητα ή την λίγη αποτελεσματικότητα ε, της Γουάντα, της Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά του ντόπινγκ και των εθνικών ε, κυβερνήσεων, ε, των εθνικών ομοσπονδιών, των διαφόρων αθλημάτων που είναι κατά του ντόπινγκ κτλ. Όπως λέμε και εμείς ε, στην μελέτη, είναι απαραίτητη η ανάλυση, όπως αυτή στην οποία θα προβεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν. Πρέπει να γίνει ανάλυση λοιπόν. Το πρόβλημα επίσης για μια δράση ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι μέχρι στιγμής οι δράσεις αυτές δεν κατάφεραν να βρουν σύμφωνα όλα τα κράτη-μέλη. Ίσως τώρα με το άρθρο 165 έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να δούμε αν τελικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμφωνήσουν ε, σε μια στρατηγική για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, γιατί υπάρχουν πολλές στρατηγικές και ετερόκλητες μεταξύ τους. Κάποιοι τιμωρούν ε, τους αθλητές, ε, σε κάποιες χώρες ενώ, κάποιοι άλλοι νόμοι όχι, σε άλλες χώρες. Πέραν λοιπόν της χρηματοδότησης στην Γουάντα, δεν υπάρχει πολιτική βαρύτητα, δεν έχει πολιτικό βάρος ε, αυτή η οργάνωση. Και τώρα δίνω το λόγο στον Ρίτσαρτ για τα υπόλοιπα. Ε, I'll try be brief. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει τη νομική βεβαιότητα. Ακούστηκαν ερωτήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς στον αθλητισμό. Το συμπέρασμά μας προκύπτει από την απόφαση με Καμεντίνα. στην οποία το ΔΕΚ είπε πως ε, καλύτερο είναι να κρίνουμε κατά περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σε διαφορετικό πλαίσιο και τίθενται ζητήματα αναλογικότητας που απαιτούν να κρυθεί ξεχωριστά η κάθε περίπτωση και ως ερευνητική ομάδα είμαστε υπέρ αυτής της προσέγγισης. Πρέπει να θυμόμαστε πως όταν εκδίδονται κατευθυντήριες γραμμές, οι κατευθυντήριες γραμμές δεν προσφέρουν νομική βεβαιότητα, μπορεί ακόμα και να περιπλέξουν τα πράγματα δεδομένου του ότι μπορεί να τις προσβάλλει κάποιος εάν ε, εκδώσει κατευθυντήρης γραμμές Κομισιόν η συνθήκη δεν ε, δίνει στην Κομισιόν την δυνατότητα βέβαίω να κάνει κάτι αντίθετο με την συνθήκη και αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο και το κρίνει σύμφωνα με την απόφαση την οποία προανέφερα. Οπότε ε, από νομική σκοπιά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εποπτεία των επιλογών που κάνουν ε, οι φορείς ε, που διοικούν, οι οποίοι είναι αρμόδιοι βεβαίως για το δικό τους το άθλημα. Και θα πρέπει βεβαίως να αναθεωρήσουν τους κανονισμούς τους ε, για να συμφωνούν με το κοινοτικό δίκαιο και μπορεί να συνεισφέρει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το διάλογο μέσω της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου επίσης και μέσω ενός πιο επισήμου δομημένου διαλόγου, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά η Κομισιόν να πάει σε ένα σύστημα θεματικού διαλόγου για συγκεκριμένα ζητήματα, για τη ρύθμιση π.χ. των μάνατζερ ή για ένα οικονομικό fair play, αλλά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και να επιδείξει μια ευελιξία η Κομισιόν που την έχει επιδείξει νομίζω π.χ. για τους μάνατζερ είναι ευαίσθητη στιγμή γιατί οι φορείς της διοίκησης του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή νομίζω εξετάζουν μια αναθεώρηση των σχετικών κανονισμών και θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους φορείς του ποδοσφαίρου να ρυθμίσουν τα του οίκου τους, στο άθλημά τους δηλαδή. Και όπως είπα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πολλά να κάνει για να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των φορέων αυτών, όπως ξεκαθαρίζει το άρθρο 165 και ε, βεβαίως για να διευκολύνει και την κατάσταση μεταξύ των διαφόρων ε, αθλημάτων και την άσκηση του Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους συντάκτες της μελέτης, ευχαριστούμε την Κομισιόν που άκουσε τα όσα υπόθηκαν και συνεισέφερε. το άρθρο 165, όπως αντιλαμβάνομαι, δεν θέλουμε να μας περιορίζει, αλλά ακόμα και αν δεν είναι η νομοθετική βάση για εναρμονισμό σε κάποιες περιπτώσεις, να δίνει μία ορμή στην ε, Κομισιό να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε κάποιους τομείς από ό,τι μέχρι τώρα. Την τελευταία σας απάντηση εγώ την ερμηνεύω ως εξή. Ε, το θέμα, παραδείγματο χάρη με τους μάνατζερ των παικτών ή το οικονομικό αυτό fair play, ως εξή λοιπόν, η Κομισιόν στο πλαίσιο του 165 μπορεί να δώσει ένα ερέθισμα στους φορείς τους αθλητικούς για να δημιουργήσουν βεβαίω τις δικές τους, τις ε, συνθήκες, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές και να βοηθήσει λοιπόν η Κομισιόν να διευρυνθεί ο κύκλος, αν θέλετε, που δεσμεύεται από αυτά τα πράγματα. Να συνεργαστεί δηλαδή η Κομισιόν με τους διαφόρους συνδέσμους, έτσι ώστε οι μηχανισμοί που έχουν βρεθεί σε κάποια αθλήματα να συμπεριλάβουν ένα μεγαλύτερο κύκλο για να υπάρξει, αν θέλετε, ένα είδος εναρμόνισης χωρίς ίσως να αναγκαστεί η Κομισιόν να νομοθετήσει με διαφορετική ε, νομική βάση. Οπότε το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο από την Κομισιόν βεβαίως ε, δεν ε, νομίζω εκεί πέρα να υπάρχουν όρια πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Υπάρχει και ο κύριος Μαυρομάτς που ήταν καιρό εδώ πέρα στην Επιτροπή μας και προσπάθησε να συνεισφέρει πολύ δημιουργικά στις προτάσεις αυτές της Κομισιόν, έτσι ώστε αυτό το οποίο επιθυμούμε εμείς και υπάρχει και στη Λευκή Βίβλο να εφαρμοστεί εν μέρη και στην πράξη. Εγώ μπορώ να πω λοιπόν πως από όλα τα διάφορα αιτήματα που έχω λάβει στο γραφείο μου από διάφορες ενώσεις, μπορώ να σας πω πως αναμένουν να κάνουμε κάτι παραπάνω από καλά λόγια. Γι' αυτό ελπίζω και η Κομισιόν να παρατήρησε σήμερα πως αναμένουμε κάποια πράγματα από εσάς, να μην καθυστερείτε τόσο όσο πρέπει να είναι βεβαίω η νομική, αλλά να προσπαθήσετε, όπως είπα, να είστε κάπως δημιουργικοί Ελπίζω να εκπροσώπησα και να εξέφρασα και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά τους συντάκτες της μελέτης, η οποία θα μας βοηθήσει και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και εμείς για να παρακινήσουμε την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τα διάφορα. Όχι. Α, έχουμε χτες την συνεδρίαση των συντονιστών τα λάβατε στο email σας, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κυρία Καμεριέβα, έχει πρόβλημα. Όχι, όχι κανένα πρόβλημα, ε, ήμουν εκεί. Να σας πω μόνο πως είχαμε κάποιες δυσκολίες, ε, γιατί ε, είχαμε κάποιους εμπειρογνώμονες για τον αθλητισμό, εάν κάποιος βεβαίως λείψει μπορούμε να τον απληρώσουμε με τους γνωστούς εμπειρογνώμονες. Ωραία, βεβαίως, αν έχετε κάποια κάποιο πρόβλημα με τους συντονιστές, όχι, ήταν σε ομοφωνία συμφωνήσαμε. Λοιπόν, τίποτα στα διάφορα, όχι. Και 15, επόμενη συνεδρίαση 26 και 27 Οκτωβρίου. 27 έχουμε την ακρόαση και σας περιμένω όλους. Όχι μόνο αυτή η πλευρά και από εδώ παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Σχολάνε και νωρίς ερμηνεία. Λοιπόν, λίγη συνεδρίαση.